Good morning everyone and... Καλή σας μέρα. Άκουσα ότι θα προσταθούν και άλλοι εδώ όσο περνάει η ώρα. Σήμερα το πρωί λοιπόν κυρίσω την άναρξη τη συνεδρίασή μα τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και καλωσορίζω εδώ και του παρατηρητέ μα, γιατί δεν έχουμε συχνά κοινό ε, στην Επιτροπή αυτή, οπότε πολύ χαιρόμαστε που σα έχουμε μαζί μας. Επίσης μεταδίδεται και στο διαδίκτυο η συνεδρίαση αυτή, οπότε υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μας ακούνε στο διαδίκτυο. Καλωσορίζω επίσης την κυρία Κένινγκ εδώ, η οποία είναι η πρόεδρος του ενιαίου Συμβούλιο Εξυγένσης και θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε ολοκληρώσει εδώ τις διοργανικές διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο όσον αφορά το πακέτο για τις τράπεζες που πρόκειται για την αναθεώρηση οδηγία για την εξυγίαση των τραπεζών, πρόκειται για την οδηγία επίσης κεφαλικών απαιτήσεων. Όλα αυτά βέβαια τα λέω με τα αρχικά τους, BRRD, CRR, αλλά όλα αυτά, πάση περιπτώσει, είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Το πακέτο για τις τράπεζες θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος για να έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα με μεγαλύτερη αντοχή. Χαίρομαι πολύ λοιπόν για αυτή την πρόοδο που ολοκληρώθηκαν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις. Επανειλημμένη ήταν εδώ η κυρία Κόνιγκ μαζί μας ξανά και ξανά και μας βοήθησε πάρα πολύ με τις απόψεις της για το θέμα. Μας βοήθησε να καταλάβουμε κάποια ζητήματα που τίθενται κάθε φορά που νομοθετούμε σε αυτό το τομέα. Την ευχαριστώ λοιπόν προσωπικά αλλά και εκ μέρους της Επιτροπής μας για την συνδρομή της όλο αυτό τον καιρό. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις μετά την αρχική της παρουσίαση. Έχετε το λόγο κυρία Κένινγκ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Επιτρέψτε μου να αρχίσω επιστρέφοντας στις ευχαριστίες, γιατί η Επιτροπή αυτή ε, πάντα διαφερόταν πολύ, έθετε πολλά ερωτήματα και προσφέρει τροφή για σκέψη και σε μας. Οπότε και εγώ σας ευχαριστώ για όλα αυτά. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η αυτή φορά είναι η 16η φορά που βρίσκομαι εδώ, σε αυτή την Επιτροπή. Και θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που ήμουν εδώ, πώς περνά ο καιρός. Λοιπόν, ε, είπατε ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ τα τελευταία αυτά πέντε χρόνια. Τον Μάιο, απλώς για να σας θυμίσω μερικά πράγματα, τον Μάιο του 2014 η Οδηγία για την Εξυγίανση Τραπεζών άρχισε να ισχύει και τον Ιούλιο του 2014 είχαμε τον ενιαίο μηχανισμό ε, εξυγίανση, τον κανονισμό για αυτό το μηχανισμό δηλαδή και στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς είχαμε και το τραπεζικό πακέτο, το οποίο συμφωνήθηκε τελικά και πραγματικά ε, περιμένω να τον εγκρίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη αυτού του μήνα. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει ε, γενικά το πεδίο πάνω στο οποίο εργαζόμαστε. Για μας είχαμε πάρα πολλή δουλειά ε, κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Εμείς βέβαια αρχίσαμε λίγο αργότερα από εσά τη θητεία μας και με επιτυχία προχωρήσαμε και μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι πάει καιρό, αλλά είναι κάτι επίκαιρο ακόμα και είναι η εξυγίανση της Banco Popular, της Ισπανικής Τράπεζας. Και νομίζω ότι σωστά θα πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση αποδείξαμε ότι το πλαίσιο το οποίο εσείς δημιουργήσατε λειτουργήσε και βοήθησε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα όχι μόνο στην Ισπανία αλλά πέρα και από αυτήν. Οπότε συνεχίζει η εξυγίανση απρόσκοπτα και δεν χρειάστηκε να πληρώσουν την ύφη οι φορολογούμενοι. Όμως πρέπει να σας πω εδώ, γιατί και αυτό το έχω συζητήσει και με τα σπανικά μέσα ενημέρωσης και αλλού, να ξέρετε ότι όταν φτάνουμε σε στάδιο εξυγίανσης, Πρόκειται για μια διαδικασία αφαιρεγκαιότητας, έτσι. Οπότε απώλειες υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν απώλειες σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποιοι λοιπόν θα χάσουν χρήματα σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό και σωστό, ότι αυτοί που θα χάσουν χρήματα είναι οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι. Αυτό έγινε και με την Banco Popular. Οπότε νομίζω ότι εδώ μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι επεξεργαστήκαμε αυτή την περίπτωση αποτελεσματικά. Εμείς δημιουργήσαμε ε, τον ε, ενιαίο, το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγένσης μετά από το αντίστοιχο Ταμείο και προσπαθήσαμε να καταφέρουμε και το, για το 2023 να έχουμε το 1% των ε, καλυμμένων αποταμιεύσεων. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι που κυρίως κάνουμε, έχουμε ασχοληθεί με την εξυγένση και τα πλαίσια εξυγένσης όλων των τραπεζών. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό για να ενισχύσουμε τα σχέδιά μας για την εξυγένση. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι η εξυγίανση και η αποτελούν την εξαίρεση. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να προχωρήσουμε στη διάλυση μιας τράπεζας, αυτό είναι σίγουρα η εξαίρεση, τις περισσότερες φορές προχωράμε στην εξυγίανση, έτσι κι έχουμε το πρώτο βήμα και μετά το δεύτερο βήμα. Πάντως, εμείς ξεκινήσαμε το 2015, την 1η Ιανουαρίου, από μηδέν προσωπικών, έχουμε σήμερα 400 υπαλλήλους πλήρης απασχόλησης. Αυτό θα είναι το νούμερο στα τέλη αυτής της χρονιάς. Ο στόχος μας επίσης σταθιακά άλλαξε. Αρχικά θέλαμε να φτιάξουμε τα πλαίσια, να εκπονήσουμε την... και να πτύξουμε μια πολιτική και τώρα προχωράμε στην εξηγένση και κοιτάμε ε, πώς θα καθοδηγήσουμε σωστά τις τράπεζες προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή το πλαίσιο αυτό της εξυγένσης. Και έχουμε συνεργαστεί στενά και με τις εθνικές αρχές αλλά και με τις ίδιες τις τράπεζες προκειμένου να αναπτύξουμε πρώτα απ' όλα τις πολιτικές μας και μετά να τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, να τελοποιήσουμε. Το είπα και την προηγούμενη φορά και υποφελούμε από κάθε ευκαιρία να το πω ότι οι τράπεζες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Εκείνες είναι υπεύθυνε προκειμένου να μπορούν να περάσουν σε εξυγένση, να έχουν ε, καλή διαχείριση και όντως οι διαχειριστικές τους ομάδες δουλεύουν πάνω σε αυτά. Το κάνουν. Το να περιμένουμε να γίνει πρώτα ζημιά και μετά να προχωρήσουμε δεν είναι λύση. Κάποιες βέβαια όταν δεν κάνουν ό,τι πρέπει εμείς τους το λέμε έχουμε τα εργαλεία που χρειαζόμαστε στη διάθεσή μας. Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει να φροντίσει τράπεζα να εξηγιανθεί. Είπαμε, δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένουμε να συμβεί η ζημιά. Εμείς θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Έχουμε το MRL, που είναι οι ελάχιστες απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων και αποδεκτών απαιτήσεων. Είναι η πιο γνωστή προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί να εξηγηθεί μια τράπεζα, εφόσον βέβαια έχει φροντίσει να έχει αρκετά κεφάλαια για να μπορεί να απορροφήσει τις απώλειες και να μπορεί να ανακεφαλαιοποιηθεί. Αντικαθιστούμε δηλαδή την χρηματοδότηση από πλευρά του φορολογούμενου, το bailout, από το bail-in. Οπότε οι ομολογίες και οι μετοχές ε, καλύπτουν τις απώλειες. Εμείς έχουμε δουλέψει σκληρά για την πολιτική μας και το έχουμε κάνει σταδιακά. Εφαρμόζουμε μία ε, πολιτή προσέγγιση στο MRL και η τελευταία μας ε, πολιτική η οποία τον Ιανουάριο δημοσιεύτηκε, ε, τονίζει την ποιότητα και την ποσότητα του MRL και εισάγει στον μηχανισμό αυτό ειδικέ απαιτήσει για το πού πρέπει να βρίσκονται τα MRL, πού είναι οι υποχρεώσει μέρε εξασφάλιση κλπ. Όλα αυτά βέβαια συνοδεύουν το τραπεζικό πακέτο και γίνονται προκειμένου να είμαστε σε θέση να περάσουμε στο δεύτερο γύρο της Οδηγίας για την Εξυγίανση Τραπεζών, το BRRD2, και έτσι να προχωρήσουμε και με την πολιτική μας για το MRL. Το επίπεδο βέβαια εξαρτάται για το πώς θα προχωρήσουμε στην εξυγίανση αλλά το MRL δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τις εργασίες μας. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο το 2017, το 2018 και τώρα έχουν αναδειχθεί τέσσερις παράγοντες. Ο ένας είναι η δομή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το άλλο είναι η διαχείρισή τους, το άλλο είναι η λειτουργική του συνέχεια και το τέταρτο είναι η επικοινωνία. Και οποιοδήποτε έχει ασχοληθεί με την οργάνωση των τραπεζών δεν εκπλήσεται που αυτά τα τέσσερα θέματα είναι βασικά για μας. Και ξεκινάω με την δομή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι κάτι πολύ σημαντικό κυρίως για τις μεγάλες τράπεζες διασυνοριακές που χαρακτηρίζονται από περίπλοκες δομές. Και αυτό έχει να κάνει με νομοθεσία κλπ. Και έτσι γίνεται πιο περίπλοκο το θέμα της εξυγίανσής τους. Όμως εδώ θα ήθελα να σκεφτούμε λιγάκι ακριβώς το MRL, δηλαδή ο τρόπο που χρηματοδοτείται μια τράπεζα είναι στοιχείο κλειδί και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν κοιτάμε την εσωτερική χρηματοδότηση των τραπεζών. Τι συμμετοχικέ επενδύσει δηλαδή, προκειμένου μια τράπεζα να μπορεί να ανταποκριθεί στο MRL. Πρέπει αυτή η χρηματοδότηση να είναι ρεαλιστική. Επίση, οι τράπεζε θα πρέπει να εισάγουν το λεγόμενο playbooks που έχουμε αντιγράψει και εμείς από την Αμερική που περιγράφει τη δομή της τράπεζας και λέει ποιο είναι το κεφάλαιο που χρειάζεται ε, προς τα κάτω και ποιο, ποιο είναι το κεφάλαιο που χρειάζεται για την απορρόφηση απολειών. Βέβαια, εύκολα το λέει κανείς, δύσκολα το κάνει. Αλλά εμείς έχουμε ξεκινήσει από αυτή την χρονιά να χρησιμοποιούμε αυτά τα playbooks για να περιγράφεται αυτή η σχέση. Και δεν είναι μόνο οι τράπεζες που πρέπει να φροντίσουν για τα playbooks, πρέπει και σε εθνικό επίπεδο να υπάρχουν εγχειρίδια από τις εθνικές αρχές, γιατί υπάρχει το διοικητικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, αφαιρεγγιότητας, όλα αυτά είναι εθνική νομοθεσία. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε στην χώρα Α, στη χώρα Β πώς λειτουργούν όλα αυτά. Έπειτα έρχομαι στα, στη διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών. Οι περισσότερες τράπεζες δεν είναι ακόμα σε θέση να πατήσουν ένα κουμπί και να μας δώσουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε προκειμένου να αποτιμήσουμε την κατάσταση ή να συγκεντρώσουμε στοιχεία για την ε, δομή των υποχρεώσεών τους και να βάλουμε σε κάποια κατηγορία τις ε, ε, υποχρεώσεις τους με κάποιε τράπεζε μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Ζητάμε από τι τράπεζε λοιπόν να φροντίσουν να μας διευκολύνουν. Έχουμε δημοσιεύσει, και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά εδώ το σώμα, το Φεβράριο που μα πέρασε, ένα πλαίσιο για την αποτίμηση. Και για κάποιον που δεν είναι τόσο κοντά στο έργο μας μπορεί να το κοιτάξει και να εκπλαγεί έχει να κάνει με εμπειρογνώμονες, δεν έχει να κάνει με τις τράπεζες, έχει να κάνει με ειδικού. Γιατί οι αποτιμήσεις που γίνονται σε περίπτωση εξυγένσης πρέπει να γίνονται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Εμείς έχουμε βάλει τις απαιτήσει μας, τις προσδοκίες μας και πάντα λέω και επανέρχομαι στα δεδομένα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προσπαθούμε να καθορίσουμε τι ακριβώς σημαίνει όσον αφορά τις προσδοκίες μας από τις τράπεζες προκειμένου να είναι σε θέση να μας δώσουν τις πληροφορίες που θέλουμε. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Οι τράπεζες πάντως μπορούν να ε, καταλάβουν και αυτές πολλά. Έπειτα έρχομαι στην ε, επιχειρησιακή συνέχεια. Δηλαδή σε περίπτωση που έχουμε μια εξυγίανση, οι συμβάσεις που έχουν οι τράπεζες με τους παρόχους υπηρεσιών να μπορούν να συνεχιστούν. Να μην φτάνουμε μια Δευτέρα πρωί δηλαδή χωρίς να έχουμε καθόλου πάροχους. Έπειτα έρχομαι στην ε, διακυβέρνηση και την επικοινωνία και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προετοιμάζεται έγκαιρα. Τώρα, έρχομαι στις προτεραιότητές μας για το 2019. Θα έλεγα ε, μία από τα ίδια. Έχουμε τις εσωτερικές μας προτεραιότητες που είναι ότι δουλεύουμε στον ε, κύκλο σχεδιασμού εξηγιάνσεων για το 2019 και ε, για τις αρχές του 2020 και οι, οι υπηρεσίες μας, οι συνεργάτες μας το έχουν ήδη πει και είναι αυτό το πιο σημαντικό ότι η κάθε τράπεζα πρέπει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας για το 2019. Που σημαίνει ότι αν δεν το κάνουν, περνάμε στο επόμενο στάδιο. Και τέλος, δουλεύουμε για να ενημερώσουμε τα δικά μας εσωτερικά εγχειρίδια και ετοιμάζουμε και ένα εξωτερικό ε, που αναφέρεται δηλαδή στις προσδοκίες που έχουμε από τις τράπεζες, τι περιμένουμε από αυτές. Αυτό θα γίνει και περιμένουμε βέβαια και την υλοποίηση του BRRD2. Και θα ολοκληρώσω με τις επιθυμίες μας. Και ποιες είναι εσείς, όσοι από εσά επανέρθετε στον επόμενο κύκλο, είναι να ολοκληρωθεί η κεφαλαιακή ένωση γιατί πρέπει όλες οι κεφαλικές αγορές να έχουν το MRL. Να εφαρμοστεί επίσης, τέλος πάντων όσο γίνεται να ολοκληρωθεί το έντις και επίσης, και με έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέω, εναρμόνιση, αν μη τι άλλο, της νομοθεσίας για την αφαιρεκαιότητα όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έτσι ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα με τη χώρα μέλος. Αυτές είναι οι ευχές μας, λοιπόν. Προς το παρόν έχουμε πάνω από 19 διαφορετικές νομοθεσίες για την αφαιρεγκαιότητα στις χώρες μέλη. Η ρευστότητα επίσης στην εξυγίαση και το backstop είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύουμε, τον μηχανισμό αυτών προστασίας δηλαδή. Γίνεται κάποια πρόοδος, περισσότερο έχουμε προχωρήσει από ό,τι στη ρευστότητα. Αυτά και τελειώνω λέγοντας ότι έχουμε διανύσει έναν μακρύ δρόμο. Έχουμε πετύχει πολλά. Οι τράπεζες είναι περισσότερο αντοχής και γερές από ότι όταν φτάσατε εδώ. Είναι καλύτερη η ποιότητα και η ποσότητα του κεφαλαίου τους. Αλλά συνεχίζουμε και στο έργο μας για να τις βοηθήσουμε να μπορούν να διασωθούν πιο εύκολα. Κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν, εσάς και τους συνεργάσεις σα και τώρα είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κένινγκ. Θα έχουμε ερωτήσεις ως εξή για πέντε λεπτά. Δηλαδή κάνετε την ερώτησή σας, μετά την απάντηση και αν δεν έχουν περάσει πέντε λεπτά σε αυτό το διάλογο μπορείτε να επανέλθετε. Με τη σειρά των πολιτικών ομάδων, πρώτα, πρώτη ερώτηση από το ΕΛΚ, ο κύριος Χόκμαρ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την ομιλία κύριε Μα Μας είπατε ότι είστε για πρώτη φορά εδώ, στο πλαίσιο δηλαδή μιας παρουσίασης των ε, υποχρεώσεων σας ε, και των όσων κάνετε στο πλαίσιο του μηχανισμού. Και εμένα είναι η τελευταία μου φορά που παρευρίσκομαι και πρέπει να πω ότι πολλά επιτεύχθηκαν ε, αυτόν τον τελευταίο αυτήν την τελευταία περίοδο και πράγματι ε, σε ό,τι αφορά και τις ε, τραπεζικές αγορές αλλά και σε ό,τι αφορά τα παράγωγα έχουμε προχωρήσει αρκετά και σε ό,τι αφορά τα capital requirements, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις σχετικές, τα σχετικά κανονιστικά πλαίσια σε ό,τι αφορά την τραπεζική ένωση έχουν όλα τους προχωρήσει. Άρα λοιπόν ε, μπορεί κανείς να πει στις αρχές εξυγίανσης τη σήμερον ημέρα ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από ποτέ γιατί ποτέ δεν είχαμε ένα τόσο ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε ακριβώς να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα εξυγίανσης με τον τρόπο που μπορούμε σήμερα. Δηλαδή πολύ συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένους κανόνες ό,τι αφορά την ιεραρχία, τα τύλα, MRL και ούτω καθεξής. Και αντιλαμβάνομαι ότι έχετε και κάποιες επιθυμίες για το μέλλον, κάποιες ευχές αν θέλετε, πράγματα που θέλουν να γίνουν, αλλά αυτή τη στιγμή ε, έχετε τα απαραίτητα εργαλεία για να επιτύχετε αυτά που καλείστε να επιτύχετε ως αρχαίος μηχανισμός. Και θα ήθελα να μας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε σε ό,τι αφορά τα σχέδια εξυγίασης που είναι απαραίτητα ε, και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο πλαίσιο αν θέλετε, έτσι ώστε να πείσουμε και τι κυβερνήσει αλλά και τι τράπεζε, ότι κατά την επόμενη κρίση τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να περάσουμε προ τι τράπεζε, προ την αγορά, προ του επενδυτέ, προ του καταναλωτέ, ότι κατά την επόμενη κρίση τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και νομίζω πω αυτό το μήνυμα θα πρέπει να έρθει από τη δική σα ε, πλευρά. Δηλαδή να πείτε τι ακριβώ θα κάνετε την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κρίση, ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Απάντηση. Ναι. Ε, στην περίπτωση της Banco Popular νομίζω προσπαθήσαμε να καταδείξουμε αυτό ακριβώς ότι δηλαδή το πλαίσιο που δημιουργήσατε πράγματι είναι το κατάλληλο. Είμαστε σε θέση δηλαδή να λάβουμε πολύ βραχή πρόθεσμα τις απαραίτητες αποφάσεις. Αυτό που πρέπει λοιπόν να περάσουμε ως μήνυμα και το οποίο ήδη αναφέρθηκε είναι ότι μία εξυγίαση είναι πάντοτε μια περίπτωση όπου μια τράπεζα έχει απολέσει χρήματα ή δεν είναι πλέον φερέγγια ή είναι σχεδόν αφαιρέγγια, δηλαδή έχει απολέσει μεγάλο τμήμα της ρευστότητάς της. Οπότε, ε, δεν είναι μια περίπτωση όπου δεν έχει υπάρξει ζημία. Δηλαδή υπάρξει, ακριβώς, υπάρχουν ζημίες οι οποίες θα πρέπει να κατανεμηθούν με έναν τρόπο και ακριβώς τις κατανέμουμε ε, με τρόπο τέτοιο στους ε, οτσιές αφορούν μόνο τους μετόχους και εκείνους που έχουν λάβει τίτλους έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε στην ίδια κατάσταση όπω εκείνη που ίσχυε πριν από το νέο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή όπου οι καταναλωτέ μέσω ακριβώ του σχεδίων διάσωσης έπρεπε να χρηματοδοτήσουν, να αναχρηματοδοτήσουν αυτέ τι τράπεζε, επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Θα πρέπει λοιπόν να εκπαιδεύσουμε, αν θέλετε, το κοινό μα ότι αν κανεί κάνει μια επένδυση σε ένα σε ένα τίτλο γενικότερα σε τράπεζε, υπάρχει ο κίνδυνο να απολέσει χρήματα. Και νομίζω πω. Και είμαι πεπισμένο ότι στο πλαίσιο των σχεδίων εξυγίανση μας και στο πλαίσιο το, το νέο πλαίσιο μάλλον νομίζω πως δημιουργούμε ακριβώς ε, ρεαλιστικό αν θέλετε, δηλαδή έτοιμο για την πραγματικότητα το νέο πλαίσιο. Και ε, σε ό,τι αφορά αυτό το θεωρητικό ερώτημα που τίθεται, ως προς το τι ακριβώς θα κάνουμε την επόμενη φορά. Ε, ελπίζουμε να μην προκύψει, αλλά αν προκύψει, τι θα πρέπει να κάνουμε, πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση, ποιες θα είναι διαφορετικές εναλλακτικέ που θα έχουμε στη διάθεσή μας και ποιε είναι οι επιπτώσεις. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό έρχεται να απαντήσει ο σχεδιασμός για την εξυγίανση. Και το γεγονό ότι δημιουργήσατε ακριβώς ένα σαφές πλαίσιο και μια σαφή ιεραρχία ανάμεσα στους διάφορους πιστωτές μας επιτρέπει σε ό,τι αφορά για τις μεγαλύτερες τράπεζες και τις απαιτήσει του πυλώνα 1 να επιτύχουμε πραγματικά μια πιο χρηστή ε, διαχείριση από την πλευρά τους. Οπότε σίγουρα ε, ε, σε περίπτωση εξυγίανσης έχουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι ελπιρό, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή το πλαίσιο είναι καλύτερο. Δεύτερη παρέμβαση, τον κύριο Χόγκμαν. ναι, Ευχαριστώ που το αναφέρετε, γιατί αυτό που θέλω να διασφαλίσω εγώ είναι ότι θα πούμε ότι, να πούμε το ότι το νομοθετικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ε, υπάρξει περαιτέρω νομοθεσία. Θα πρέπει να εφαρμοστεί πλέον με τον σωστό τρόπο. Και αυτό λοιπόν είναι που απαιτείται αυτή τη στιγμή. Να έχουμε ακριβώ αυτή την κοινή κατανόηση ότι πραγματικά έχουμε δημιουργήσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που χρειαζόμαστε. Ναι. Ναι, ο κύριο Σόγκμακ. Ε, ναι, και αυτό που είπα μόλις τώρα ήταν μία δήλωση, δεν έθεσα ερώτημα. Κύριε Πέρας, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε, κύριε πολύ την κυρία Κιόνιγκ. Ε, είναι η τελευταία ανταλλαγή θέσεων και πρέπει να πω ότι με την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών τα τελευταία χρόνια είχαμε πάρα πολύ καλή και επικοδομητική συνεργασία. Δύο ερωτήσει. Πρώτον, είπατε στην ε, επιστολή ευχών και επιθυμιών ε, ότι ε, χρειάζεται η Κεφαλιακή Ένωση για την ενίσχυση της ρευστότητας των αγορών. Γνωρίζετε ίσως ότι ήμουν η συγγήτρια για το θέμα της αναθεώρησης των εποπτικών αρχών. Όσο τα, τα κράτη-μέλη δεν δέχονται έναν πραγματικό ευρωπαϊκό μηχανισμό επιτήρησης των κεφαλαιακών αγορών, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα επιτύχετε αυτήν την κεφαλαική ε, ένωση. Ε, και ε, βεβαίως υπάρχουν χώρες, μία εκ των οποίων γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, που δεν θέλουν και πάντα βρίσκεται σε αντιπαράθεση και σε αντίθεση με τη συζήτηση αυτή για το θέμα της Κεφαλαϊκής Ένωσης και επομένως νομίζω ότι εάν ε, καταφέρουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω από τα εθνικά ζητήματα θα μπορέσουμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε μια ιταλική περίπτωση. Είναι ε, η περίπτωση του Τέρκα της Ιταλίας όπου θεωρήθηκε ότι μια και πρόκειται για ένα ε, ε, φαντ το οποίο, το οποίο ελέγχεται από το δημόσιο δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Αυτό ίσως κόστησε και τις εκλογές σε ένα συγκεκριμένο κόμμα στην Ιταλία. Σκέφτεστε μήπως, θεωρείτε μήπως ότι θα έπρεπε να είχατε κινητοποιηθεί εσείς από την αρχή και πιο ξεκάθαρα όσον αφορά την δυνατότητα της προηγούμενης Ιταλικής κυβέρνησης ε, να χρησιμοποιήσει αυτό το, ε, αυτό το ταμείο απάντηση της κυρίας Κιονίκα. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι η, ε, αγορά η Ένωση της Αγοράς Κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω γιατί ε, το, ε, το διαπιστώνουμε και όταν μιλάμε για το MRL και οι τράπεζες λένε ότι ναι, αυτό αποτελεί πρόκληση στην Ευρώπη και κυρίως όσον αφορά την Ένωση Κεφαλαίων αγορών ε, και ε, ε, βεβαίως εδώ πρέπει να αναφέρουμε και τη χώρα η οποία ενδεχομένως θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Το δεύτερο θέμα το οποίο αναφέρεται είναι αυτό το Ταμείο Τέρκα, το οποίο αφορά μια μικρή Ιταλική τράπεζα η οποία κατέρευσε αν ε, θυμάμαι καλά το 12 ή το 13 δηλαδή πολύ πριν ε, δημιουργηθεί η Τραπεζική Ένωση. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση ε, το πρόγραμμα εξασφάλισης καταθέσεων της Ιταλίας χρησιμοποιήθηκε και βεβαίως εγώ δεν θέλω να σχολιάσω το θέμα αυτό γιατί συνέβη πριν από τη δημιουργία του πλαισίου μας ε, και δεν ασχοληθήκαμε εμείς Ωστόσο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ενδεχομένως μπορεί να μας βοηθήσει αυτή η συζήτηση για να ξαναζωντανέψουμε κατά κάποιο τρόπο τη συζήτηση περί το έντισε, καθώς επίσης και τη συζήτηση για το τι ακριβώς, ποιος ακριβώς θα πρέπει να είναι ο ρόλος ενός μηχανισμού εγγύησης καταθέσεων. Υπάρχει βέβαια και η οδηγία που αποτελεί το βασικό ε, μοντέλο, δηλαδή πληρωμή μετά από 7 ε, μέρες επανειλημμένα θα με έχετε ακούσει να λέω ότι κάποια εναλλακτικά μέτρα όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφερθούν επιχειρήσεις κάτω από την ομπρέλα άλλων αρχών, ότι τα εναλλακτικά μέτρα θα έπρεπε να εφαρμόζονται από όλες τις χώρες. Και βέβαια το κεντρικό σημείο θα πρέπει να είναι ε, το μικρότερο δυνατό κόστος και ευελπιστώ ότι αυτή η περίπτωση, οποιαδήποτε και αν είναι η έκβαση, γιατί βρίσκεται ακόμα στο πρώτο επίπεδο, ε, θα ξεκινήσει τουλάχιστον λόγω αυτού συζήτηση σχετικά με το τι ακριβώς χρειάζεται η Ευρώπη και οπωσδήποτε ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα DGS στην ε, Ευρώπη. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη όσον αφορά το, και το επόμενο πλέον κοινοβούλιο. Νομίζω ότι τώρα έφτασε η ώρα που όλοι λένε είναι η τελευταία μας συνεδρίαση. Ναι, φαντάζομαι ότι ό,τι λέμε ασχύει για το επόμενο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Κιόνικ και εξ ονόματος του ECR θα μιλήσω κι εγώ και πράγματι εμένα θα είναι η δικιά μου η τελευταία ε, συνεδρίαση. Είμαι εδώ 10 χρόνια και σκέφτομαι τι έχουμε πει και τι έχουμε κάνει εδώ σε αυτήν την Επιτροπή και τι, πόσα πολλά είχε κάνει και η δικιά σας ομάδα από την αρχή της ε, χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης ε, στην αρχή της θητείας του 2009 ήδη μας απασχολούσαν όλα αυτά τα προβλήματα, τα τραπεζικά, τα οποία μας απασχόλησαν για δύο ολόκληρες θητείες. Πολλά έγιναν, αλλά πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν και νομίζω ότι έχουμε χάσει κάποιες ευκαιρίες ε, όπως ε, ανέφερε και με συγκεκριμένη περίπτωση η κυρία Μπερέση. Ίσως θα ήθελα να ακούσω κάποια σχόλια από σας. Ε, ήδη το θίξατε κάπως το θέμα αυτό όσον αφορά όσον αφορά το λεγό, τους φραγμούς Τζοβανίνη, Τζοβανίνη Barriers, από, το, αυτό που είπε δηλαδή ο καθηγητής Τζοβανίνη και την ανάγκη εναρμόνισης τουλάχιστον όσον αφορά τα κομμάτια τα οποία αφορούν ε, τους ε, τίτλους ε, και την κεφαλιακή αγορά έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε εργαλεία τα οποία θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς μας είπατε δύο λόγια ή μάλλον τι μπορείτε να μας πείτε σχετικά με το αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν οι συνάδελφοι στο επόμενο κοινοβούλιο. Και μια και σας έχω εδώ δίπλα μου, θα ήθελα ε, να αναφερθώ και σε... στο θέμα that needed to be Όσον αφορά το θέμα των αντισυμβαλωμένων, ε, αυτό είναι δουλειά που έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Ε, νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο ισχύει στις μεγαλύτερες τράπεζες ε, και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να ολοκληρωθεί η νομοθεσία. Έχετε κάποιες ιδέες να μας πείτε σχετικά με το πώς και σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να προχωρήσουμε. Και κι, άλλο, κι άλλος αποχαιρετιστήριος λόγος, τι κρίμα όσον αφορά την αφαιρεγγιότητα, όσον αφορά την τιτλοποίηση. Νομίζω ότι αυτά είναι εργασία τα οποία ε, οδηγούν μακροπρόθεσμα στην Ένωση και, ε, Κεφαλαιαγορών. Και ε, ε βεβαίως στην ουσία είναι πολύ απλό να, να πει κανείς ότι θα πρέπει να υπάρχει ολοκλήρωση αλλά ε, ακόμα έχει αρκετό δρόμο ε, η διαδικασία κυρίως από την πλευρά των επενδυτών ε, γιατί δεν είναι το ίδιο για τον εκδότη που είναι το μικρότερο κομμάτι και η μικρότερη διαδρομή κατά κάποιο τρόπο τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από την πλευρά του επενδυτή και ποιες είναι οι ανάγκες του επενδυτή. Αναφερθήκατε εσείς στο ε, πλαίσιο, ευρωπαϊκό πλαίσιο εφερεγγιότητας. Ε, ε, ποτέ δεν είχαμε τόσο μεγάλο βαθμό φιλοδοξίας. Τώρα έχουμε ένα καλό πλαίσιο και βεβαίως το θέμα της ασφάλειας των τίτλων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν αυτό θα ολοκληρωθεί ακριβώς στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ίσως και λίγο αργότερα αργότερα Πάντως πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση γιατί διαφορετικά θα έχουμε κατακαιρματισμένη αγορά κεφαλαίων ε, και δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώσουμε την ε, ε, αγορά με αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο σημείο, έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά μέτωπα εδώ στην Ευρώπη αλλά έχουμε και το Financial Stability Board να πω ότι δεν κάναμε την πρόοδο την οποία θα θέλαμε και το FSB έκανε μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την μεγαλύτερη ασφάλεια των κεφαλαίων τη μεγαλύτερη ασφάλεια των τραπεζών, αλλά υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις ε, οι οποίες μπορεί να έχουν πρόβλημα ε, και μικρές τράπεζες που μπορεί να έχουν πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό ε, στο σύστημα είναι ότι όπως είδαμε και στις αλλαγές FSB, οι μεγαλύτερες τράπεζες, όχι μόνο οι ευρωπαϊκές αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, ε, μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα και αν κάποια από αυτές τις τράπεζες αποτύχει τότε προκύπτει πραγματικά ε, ζήτημα ε, γιατί θα υπάρχει ένα εφεντόμινο ε, και στις άλλες τράπεζες οι οποίες μπορεί να διαπιστώσουν απώλειες. Επομένως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να περιγράφουμε το πρόβλημα και Μπορούμε να το κάνουμε γιατί ε, έχουμε δυνατότητες πολλές όσον αφορά τον έλεγχο κινδύνου. Έχουμε δυνατότητες και πολύ καλά προγράμματα όσον αφορά τις δοκιμές αντοχής ε, ε, και επομένως θα πρέπει να προχωρήσουμε. και ίσως αυτό είναι και το τρίτο τμήμα της ε, ε, λύσης ε, επιτήρησης γιατί σε αυτή την περίπτωση η επιτήρηση θα, δεν θα πρέπει να είναι καθαρά εθνική αλλά να έχει διεθνή διάσταση. Εντάξει, δεν είναι δικά μου θέματα αυτά, αλλά νομίζω ότι ε, πρέπει να τα βλέπουμε πιο γενικά και όχι μόνο καθαρά εθνικά και στην εθνικά πλαίσια τα θέματα. Ναι, ναι, όχι. Είναι σίγουρα και δικιά σας δουλειά και οπωσδήποτε αυτά θα τα μεταφέρουμε στους συναδέλφου τη Επόμενη θητείας. Κυρία Κιόνεγε, θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για το γεγονός ότι ε, πραγματικά καταφέρατε σε μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσετε μια νέα οργάνωση ε, για να, την, ε, να της επιτρέψετε να λειτουργήσει εύρυθμα. Και βέβαια το γεγονός ότι έχουμε ε, πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αποσιάζουν σήμερα με την εξαίρεση του Σβέν Γκίγκολ και άλλων συναδέλφων ε, ε, οφείλεται στο γεγονό ότι ακριβώς βρίσκονται σε προεκλογική εκστατεία και δεν συμμετάσχουν περαιτέρω στι εργασίε αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Του ευχόμαστε βέβαια και καλή επιτυχία. Ε, Τώρα, ε, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά την Κάρι Τζέσ που εδρεύει στην ε, Γένοβα και την ε, Norddeutsche Landesbank. Το γεγονό ότι έχετε ακόμα πολλά που μπορείτε να επιτύχετε από την πλευρά του SRB αναφέρθηκε ήδη και από τη συνάδελφο Περμαν Πέρε. Πάντω, εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι για να αντιμετωπίσουμε τα υπολοιπόμενα προβλήματα θα χρειαστούμε δυστυχώς μία ακόμα χρηματοπιστωτική κρίση. Ε, σε ό,τι αφορά πάντως τις δύο αυτές τράπεζες που σας ανέφερα. γνωρίζουμε ε, πως ε, συμβαίνει κάτι για παράδειγμα στην Westdeutsche Handelsbank και ούτω καθεξής, μόνο όταν έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο ή αν έχει ασκήσει τρομακτικές πιέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα σε σχέση με αυτές τις δύο τράπεζες που σας αναφέρω, θα ήθελα να αναλυφθεί δράση και πάλι. Γιατί ουσιαστικά η λύση η οποία επιδιώκεται τώρα από την Norddeutsche ε, Handelsbank είναι ουσιαστικά ε, ε, το να καταλήξει σε μια συμφωνία και με τους επενδυτές οι οποίοι κατά το ίμιση είναι δημόσιοι. Όμως αυτή η λύση πραγματικά δεν είναι πλήρης. Είναι μερική μόνο και δεν βλέπω να αναλαμβάνετε δράση από την δική σας πλευρά. Οπότε θεωρώ πως ακόμα και μια τέτοια τράπεζα όπως η Norddeutsche Handelsbank θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες οι οποίοι ε, ισχύουν σήμερα στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να τοποθετηθείτε σχετικά κυρία Κόνη. Νομίζω πως ε, το γνωρίζετε όλοι και απαντώ στα αγγλικά για να μπορούν να με ακούσουν και οι υπόλοιποι πιο εύκολα. Νομίζω πως όλοι γνωρίζετε ότι η πολιτική μας είναι να μην σχολιάζουμε επιμέρους τράπεζας. Η Καρίτε είναι ένας σημαντικός ε, τραπεζικός 20 που εδρεύει στη Γενόβα, ενώ η Norddeutsche Handelsbank είναι μια σημαντική περιφερειακή τράπεζα η οποία έχει την έδρα στο ανώβερο της Γερμανίας. Και στις δύο λοιπόν αυτές περιπτώσεις ε, θα ήθελα να σε εξηγήσω λίγο την, το ρόλο που παίζει το SRB ο μηχανισμός. Όταν λοιπόν θεωρείται πως μια τράπεζα ε, βρίσκεται κοντά στο να ε, καταστεί ή είναι ήδη αφαιρέντια ε, δηλαδή με βάση και την αξιολόγηση από την πλευρά του επόπτη, του SSM, ε, που εδρεύει στη Φραγκφούρτη, και αυτό μπορεί να αποφασιστεί όμω και από εμά, με βάση δηλαδή μια σειρά από κριτήρια. Εφόσον λοιπόν υπάρξει αυτή η αξιολόγηση, ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην αφαιρεγκαιότητα ή είναι αφαιρέντια, πρέπει να αξιολογήσουμε το κατά πόσο υπάρχει δημόσιο συμφέρον για την τη αυτή τη τράπεζα ή αν αντιθέτω την αφήνουμε να ακολουθήσει την κανονική διαδικασία αφαιρετιότητε. Άρα λοιπόν να αξιολογούμε το δημόσιο συμφέρον λαμβάνοντα υπόψη δύο ειδικότερου παράγοντε. Χρηματοπιστωτική ε, σταθερότητα και κρίσιμε λειτουργίε για την εύρυθμη λειτουργία ε, της, του οικονομικού συστήματο του συγκεκριμένου κράτου μέλου και του συνόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο λοιπόν εφόσον ισχύουν αυτοί οι δύο παράγοντε ω κριτήρια κρίνουμε πως υπάρχει δημόσιο συμφέρον. Ε, και ακριβώς αυτή την αξιολόγηση κάναμε και σε σχέση με αυτές τις δύο ε, τράπεζες. Οπότε θα περιοριστώ μόνο σε αυτό το σχόλιο, δεν θα πω κάτι άλλο. Πρόεδρος, δεν ξέρω αν ε, θέλετε να σχολιάσετε και πάλι συνάδελφε. Πάντως σε κάθε περίπτωση γνωρίζετε πως όταν υπάρχει μια διαδικασία η οποία τρέχει και ονομάζονται πολύ συγκεκριμένε τράπεζε είναι πολύ δύσκολο το SRB να σχολιάσει. Ο κύριος Γκίγκολ, το λόγο για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ να προσθέσω κάτι. Πρώτα απ' όλα, δεν έχω πιστεί ότι είναι η τελευταία φορά που σας έχουμε εδώ. Τόσο το καλύτερο βέβαια για μένα και όλοι το ελπίζουμε αυτό. Δεύτερον, στη γερμανική πολιτική υπάρχει κάτι που ονομάζεται η διασύνδεση του ανώβερου. Connection. Έχουμε εδώ από την κάτω Σαξονία κάποιον και ακόμα και αν λέω ότι είναι από το Oldenburg και όχι από τον Όβερο, τόσο πάντων λέω ότι δεν μετράει. Έχουμε όμως την κυρία Κιόνινγκ εδώ και εγώ που έχω ένα e-level από το Όβερο που είναι ε, το μέρος όπου βρίσκεται και η οργάνωση αυτή, αλλά βέβαια έχουμε και τον Κλίμ εδώ που είναι από τη Βιέννη. Διαμαρτυρίες από τον κύριο Κλίμ. Εκτό μικροφώνου. ωραία. Και τέσσερι είναι από τα Νόβερο, λοιπόν. Ε, και να και τελικά αυτό γίνεται με τη γερμανική πολιτική. Οπότε η ερώτηση μου είναι για τον ε, SRB. Εσείς πιστεύετε ότι σας δυσκολεύει λίγο αυτή η υπόθεση, επειδή ακριβώς είναι στην πόλη σας, επειδή ξέρουμε ότι είναι μικροί, ξέρουμε ότι όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό το Annover Connection είναι λίγο τρομακτικό αυτή η διασύνδεση του Ανόβερου, η κλίκα του Ανόβερου. Και έρχομαι και στην ερώτηση του κύριου Κλίμ. Αν δύο μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδιαφέρονται να συγχωνευθούν, ας το πω έτσι. Και έχετε δύο αδύναμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συνήθως κοστίζει χρήματα μια συγχώνευση. Οπότε ρωτάω, εσεί λέτε δεν μπορείτε να σχολιάσετε για εξατομικευμένες περιπτώσεις. Ναι, αλλά για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, κοιτάτε αυτές τις περιπτώσεις αν έχουν βάλει χρήματα στην πάντα και εξετάζεται και το χειρότερο σενάριο ως αποτέλεσμα. Θα ήταν ε, ένας καλός τρόπος διαχείρισης, σοφρών να είσαστε σίγουροι ότι ε, τα ιδρύματα αυτά είναι καλά προετοιμασμένα. Όλους μας απασχολεί το τι γίνεται εκεί, ιδίω όταν είχαμε την τελευταία κρόση με την Deutsche Bank εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν απάντησαν σε καμία σχετική ερώτηση. Φαίνεται να είναι ισχυρή τράπεζα, αλλά μήπως δεν είναι. Οπότε γι' αυτό με ενδιαφέρει να ξέρω τι έχετε κάνει και αν έχετε προετοιμαστεί ικανοποιητικά. Η ε, κυρία Κανίγκ, να απαντήσω πρώτα για την κλίκα του Ανόβερου. Όπω ξέρετε, δεν γεννήθηκα εκεί. Εντάξει, ζω στο Ανόβερο. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει εδώ να είμαστε ξεκάθαροι. Εσωτερικά, για κάθε τράπεζα ελέγχουμε αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για μας, για το προσωπικό μας. Και ποτέ δεν είπαμε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εφόσον ζει στην ίδια πόλη. Αν υπάρχει όμως το παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Δηλαδή εσείς είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εδώ. Απάντηση. Όχι, θεωρώ πως ε, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων αν ε, έχω κάποια συναισθήματα. Δεν έχω για το ένα ή το άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανάλογα με το σε ποια πόλη βρίσκεται. Όχι. Δεν έχω καμία προσωπική σχέση ούτε με το ένα ούτε με το άλλο ίδρυμα. Το ότι είμαι από τη Γερμανία δεν σημαίνει ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων δικών μου για, όλο, για όλες τις τράπεζες της Γερμανίας, το ίδιο για τους συναδέρφους μου. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη ερώτησή σας είναι μια πολύ καλή για τις συγχωνεύσεις. Δεν είμαστε εντελώ ελεύθεροι για τον τρόπο ή για την αίσθηση που έχουμε και όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση νομίζω ότι ακριβώ υπάρχει αίσθηση ότι υπάρχουν τράπεζες που είναι αδύναμες σε ολόκληρη την Ευρώπη ισχύει αυτό και ότι η λύση είναι η συγχώνευση. Εγώ όμως πάντα έλεγα ότι η συγχώνευση μπορεί να είναι η λύση μόνο εφόσον υπάρχει μια πραγματική business ε, που έχει νόημα και στο τέλος έχουμε μια πιο ισχυρή ε, τράπεζα. Όταν έχουμε συγχωνεύσεις μεγάλων τραπεζών σκεφτόμαστε αμέσως το περίφημο too big to fail. Αλλά μην ε, βασιζόμαστε μόνο στον ισολογισμό τους μπορεί να σημαίνει ότι είναι και πολύ περίπλοκες για να αποτύχουν. Για να είμαστε τώρα πιο συγκεκριμένοι. Σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης, και το είδαμε αυτό και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, εμείς παρακολουθούμε τα πράγματα με τον εξή άξονα. Όταν έχουν συγχωνευτεί αυτές οι τράπεζες θα είναι πιο εύκολο να διασωθούν. Ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν. Αυτά παρακολουθώ. Πρώτα προσπαθώ να καταλάβω το business case και μετά να δω τι επίπτωση θα έχει η συγχώνευση αυτή. Τώρα για να απαντήσω σε μια άλλη ερώτηση που την ακούω και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρουμε λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν σχέδια εξυγένσης. Πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ποια είναι η οργάνωση των τραπεζών όταν αλλάζουν οι τράπεζες πρέπει και εμείς να ενημερώνουμε τα σχέδιά μας εξηγένσεις. Ελπίζω να είναι αρκετά αυτά που σας απάντησα. Πρόεδρος, δεν βλέπω κανέναν από την ΚΟΥ Με εκ μέρους του EFDD, ο κύριος Βάλλη. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις στην κυρία Κιόνινγκ. Η πρώτη αφορά την αναθεώρηση που θα ψηφίσουμε ε, σύντομα ε, για την ε, Τράπεζα Ανασυγκρότησης όπου αναφέρεται, όπου γίνεται αναφορά στα, ε, στις ελάχιστες απαιτήσει και τα MRL που θα ισχύσουν το 22 και το 24. Επίσης, ποσοτικές μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχουν τα MRL ε, στις διάφορες χώρες ε, και στους διάφορους τύπους τραπεζών έχουν γίνει, ε, γιατί οι συζητήσεις πολλές έχουν γίνει σε τραπεζικά περιβάλλοντα και προέκυψε ακριβώς αυτό το θέμα της αναλογικότητας ή στην εφαρμογή, γιατί υπάρχουν διάφορα πρότυπα, διάφοροι τύποι τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις από αυτών θα είναι διαφορετικές του ιδίου μοντέλου. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω αν έχουν γίνει τέτοιες ποσοτικές μελέτες και γενικότερα τέτοιες μελέτες έτσι ώστε να ε, μετρηθεί ο αντίκτυπος ε, ε, του MRL. Επίσης, σε σχέση με την απάντηση που δώσατε στον κύριο Γκίγκολ σχετικά με τις συγχωνεύσεις αυτών των τραπεζών του Big to Fail, μεγάλη συζήτηση γίνεται στα όσα λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή μεταξύ της Deutsche Bank και της Commerzbank, αλλά και γενικότερα τι γίνεται όταν δύο γίγαντες, ας πούμε, οι δύο τράπεζες τράπεζες τέτοιου ε, μεγέθους ε, συνενώνονται, ποιες είναι, ποια είναι τα μέτρα τα οποία ε, παίρνετε εσείς έτσι ώστε να αποσοβηθούν οι απειλές επί του συστήματος. Θα προσπαθήσω να απαντήσω την πρώτη σας ερώτηση. Έχετε δίκιο. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε την BRD2 που θα και βεβαίως πιστεύω ότι Μέχρι το 22 ε, ε, ελπίζουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της ε, διαδικασίας. Δεν έχει ξεκινήσει βεβαίως το BRD2 σε πλήρη ολοκλήρωση από των τραπεζών και η αξιολόγηση που κάναμε αφορούσε την στρατηγική MRL του 2018 και εκεί διαπιστώσαμε ότι για όλες τις ότι 170 δις ε, ήταν ο αντίκτυπος για τις τράπεζες ε, και αυτή τη στιγμή έχουμε 60 δις περίπου σε παράγωγα ή τέτοιου είδους ε, εργαλεία. Πιστεύουμε ότι στο BRD2 ο αριθμός των subordinated instruments θα είναι κάπως ευρύτερος αλλά θα έχουμε και τα επόμενα χρόνια ε, και γι' αυτό ακριβώς ε, είχαμε ζητήσει ήδη το 2016 και το 2017 αλλά και ξανά το 2017 είχαμε ζητήσει, 8, είχαμε ζητήσει λέω από όλε τις ε, τράπεζες να δουν πώς πηγαίνουν τα ημέρα. Δεν είναι ένας ε, κοιτάξτε, δεν είναι πολύ δύσκολος ο υπολογισμός, πάντως λέμε ότι οι τράπεζες όταν το επιτρέπουν οι αγορές ε, θα πρέπει να ξεκινούν στην έκδοση τέτοιων ε, προϊόντων και όχι να περιμένουν την τελευταία στιγμή αυτό που κάναμε είναι ότι προσέξαμε ιδιαίτερα ε, όλες ε, οι τράπεζες ε, να προσέξουν ιδιαίτερα και τις, τα MRL και τα ενδεχόμενα προβλήματα ή ελλείψεις Ε, έτσι ώστε οι τράπεζες ε, οι οποίες έχουν προβλήματα μέσα σε μία περίοδο ε, τεσσάρων το πολύ ετών να διορθωθούν. Ναι, βεβαίως γίνεται μία προσπάθεια αναλογικότητας. Αυτή είναι και η γενικότερη σκέψη μας. Ελπίζω ότι εν μέρη τουλάχιστον απήντησα στην πρώτη σας ερώτηση. Όσον αφορά τώρα τις συγχωνεύσεις όλες, ε, οποιαδήποτε ανάγκη θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί από τον επιτηρητή, ε, αυτόν δηλαδή που παρακολουθεί στενά την κατάσταση από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη μέρα ε, και υπάρχει και ο σέμα για τις μεγάλες τράπεζες που θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσει το πράσινο φως για οποιοδήποτε μέτρο. Και άλλωστε προσπάθησα να σας το πω και από την αρχή, ε, θα πρέπει να δούμε από την αρχή ποια είναι η επιχειρηματική ε, λογική και προς τα πού πηγαίνουμε. Το δεύτερο που κάνουμε είναι στην ουσία κάτι το οποίο έχει ήδη αποδειχθεί σωστό και σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δηλαδή λέμε ε, ότι επισήμως εμείς δεν έχουμε λόγο σε αυτήν την διαδικασία, δεν μπορούμε να πούμε κάτι αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε καλές σχέσεις με τους ε, επιμέρους ε, μηχανισμούς επιτήρησης. Δεν έχουμε Ε, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι ε, εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε θα πρέπει να αλλάξετε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα γιατί διαφορετικά δεν θα ε, έχετε το πράσινο φως όσον αφορά και την ρευστότητα ή την φερεγγιότητα. Στα τέλη του προηγούμενου χρόνου ενδεχομένως θα πήρε το μάτι σας ένα έγγραφο το οποίο εμείς ε, δημοσιεύσαμε σε σχέση με το Brexit. Είναι κακιά λέξη αλλά πρέπει να την πω και αναφερθήκαμε στο, στο τι περιμένουμε όσον αφορά ε, την φερεγγιότητα από πλευράς των ευρωπαϊκών ε, επιχειρήσεων. Βεβαίως εμείς ε, ε, ε, συνεργαζόμαστε πολύ με τον SSM στην Φραγκφούρτη έτσι ώστε να ξέρουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως θα μετακινηθούν προς την Ευρώπη τι ακριβώς ζητάμε, τι ακριβώς απαιτούμε. Κοιτάξτε, ε, όπως και σε ένα γάμο, ε, όταν παντρεύεσαι δεν σκέφτεσαι ακριβώς τι θα γίνει αν πεθάνεις, ε, έτσι και σε μια συγχώνευση. Όμως όλα λαμβάνονται υπόψη. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλο από το ΙΕΝΕΦ, e επομένως ξαναρχίζουμε το γύρο των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, καταρχήν θα ήθελα να εμ απορρίψω κατηγορηματικά αυτό που αναφέρθηκε ότι ε, εγώ έχω κάποιο είδος αυτής της, της, ε, της σχέσης με το ανώβερο. Εμείς μάλιστα θα πρέπει να πω ότι το 1946 κατά το πλαίσιο της ε, διοικητικής ανασυγκρότησης που είχε γίνει είχαμε αυθαίρετα ενταχθεί από την πλευρά της δικής μου πόλης στην ευρύτερη περιοχή του ανώβερου, πράγμα με το οποίο δεν συμφωνώ. Μετά, ε, κάτι ακόμα που έθεσαν ως ερώτημα συνάδελφοι ε, και ε, είναι ένα ερώτημα που απασχολεί και εμένα, αλλά θα ήθελα να το αναδιατυπώσω με πιο διπλωματικό τρόπο. έτσι ώστε να ανταποκριθώ και το δικό σα αίτημα κυρία Κιόνιχ, να μην αναφέρουμε δηλαδή πολύ συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ε, από τότε λοιπόν που έλαβε χώρα η τραπεζική και χρηματοπιστωτική κρίση, λάβαμε μία σειρά από μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την σταθερότητα του συνόλου του οικονομικού συστήματο και νομίζω πω πραγματικά δημιουργήσαμε τα κατάλληλα εργαλεία και του μηχανισμού για να το επιτύχουμε αυτό. Και να ανταποκριθούμε ακριβώ αυτή την πρόκληση. Όταν Υπάρχει λοιπόν ένα παίκτη τη τραπεζική ε, και χρηματοπιστωτική αγορά, αντιμετωπίζει λοιπόν προβλήματα όταν βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Συχνά υπάρχει ακριβώ αυτό το κάλεσμα να αναλάβει δράση το κράτο προκειμένου να μετριάζει τι αντικέ επιπτώσει. Έχουμε τώρα τον ενιαίο λοιπόν μηχανισμό ο οποίο επιτρέπει ακριβώς ε, την ε, την, την, ε, το να προβλέπετε μια ενιαία, μια τακτική διαδικασία, αν θέλετε, σε αυτών των ε, ε, τραπεζών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά, σε τέτοιου είδου σε προβληματικές περιπτώσεις, όταν αντιμετωπίζουμε μια τέτοια ένα τέτοιο πρόβλημα. Συνήθως λοιπόν αποφασίζουμε να διασώσουμε την ελόγω τράπεζα. Και εκεί βέβαια η τράπεζα, ο μηχανισμό, το δικαστήριο, όλοι του θέτουν συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένε απαιτήσει ω προ το αν ε, έχει νόημα πράγματι να διασωθεί εν λόγω τράπεζα. Παρόλα αυτά όμω, θεωρώ πω υπάρχει μια γενικότερη δυσαρέσκεια όταν ακριβώς διασώζεται με αυτόν τον τρόπο μια τέτοια τράπεζα. Οπότε θα ήθελα να θέσω το ερώτημα. Ε, τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει μέχρι στιγμής επαρκούν ή αν θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές εδώ, κάποιες ρυθμίσεις ώστε πραγματικά να ε, λειτουργήσει καλύτερο το σύστημα. Εσείς δηλαδή ω επικεφαλής ε, του ΕΣΑΠΗ, θα θέλατε... Ε, να ληφθούν περαιτέρω μέτρα έτσι ώστε να είμαστε πιο προσεκτικοί να λαμβάνουμε τις καλύτερες αποφάσεις σε ό,τι αφορά το κατά πόσο θα υπάρξει μια διάσωση ή όχι. Σε ό,τι αφορά ε, την ε, συμπερίληψη της, και της κολονίας στην πρόσης Land Province, έτσι, δηλαδή αυτά τα ζητήματα, αν θέλετε, διοικητικής ένταξης ορισμένων πόλεων, εντάξει, πραγματικά θίγομαι και εγώ από κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δημιουργήσαμε λοιπόν το και το μηχανισμό εξυγένσης και πρόκειται για μια πολιτική δέσμευση όταν λέμε ότι προβλέπουμε μια διαδικασία εξυγίανσης έτσι ώστε οι τράπεζες να είναι δυνατόν να, ε, απο, να, να, κλείσουν, θέλετε, να φαλυρίσουν, το εισαγωγικό, να πτωχεύσουν όπως οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Αλλά δεν είναι δυνατόν από τη μία προς την άλλη μέρα να πούμε ότι τα πάντα έχουν αλλάξει και ότι υπάρχει ε, μια καινούργια κατάσταση. Είδαμε το τι συνέβη και στην περίπτωση της Banco Popular. Είδαμε δηλαδή στην αρχή όπου είχαμε κάποιες περιπτώσεις ε, τραπεζών όπου τα πράγματα ήδη βρίσκονταν σε φάση αν θέλετε επίλυσης ήδη προτού τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο. Άρα λοιπόν ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από πριν. Και από εκεί και μετά βρισκόμαστε σε μια φάση εκπαίδευση εντό εισαγωγικών όλων. Ε, ε, δηλαδή παιδεία. ότι δηλαδή όταν κανείς επενδύει σε μια τράπεζα θα πρέπει να ε, μην έχει την αίσθηση ότι είναι απόλυτα εξασφαλισμένη η μία επένδυση, ότι είναι απόλυτα σίγουρη, απόλυτα σιγανή μία επένδυση σε μία τράπεζα ή τόσο στεγανή εν λόγω επένδυση όπως για παράδειγμα σε μία εξασφαλισμένη κατάθεση. Αυτό λοιπόν να το πιστεύει κανείς ή ε, πιστεύει σε ανοησίες ή δεν έχει ακριβώς λάβει την κατάλληλη ενημέρωση, δεν γνωρίζει το τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να υπάρξει αυτή η αλλαγή της νοοτροπίας, αλλά από εκεί και μετά υπάρχει το, η αίσθηση ότι δηλαδή όταν συμβεί κάτι σε μια τράπεζα ε, κατευθείαν το κράτος ε, ε, ενεργοποιείται για να διαθρώσει. Αν όμω υπάρξει για παράδειγμα ένα πρόβλημα σε μια επιχείρηση λιανικής ή για παράδειγμα σε μια μηχανολογική επιχείρηση κανένα δεν κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να, δώσουμε, να εξηγήσουμε ότι εάν πάει κάτι λάθος με μια τράπεζα εκείνοι ακριβώ που έχουν συμμετοχές, μετοχικές ή αλλε στα κεφάλαια τη τραπεζα είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να τη βοηθήσουν. Ε, για, την, για το S&D, ε, Dr. Βίντε. Ευχαριστώ. Προτού θέσω το ερώτημά μου, και εγώ σε Γερμανίδα ε, βουλευτής, να αναφερθώ στο ζήτημα της κάτω Σαξονίας. Εγώ εκπροσωπώ εδώ τη Θουριγκία η οποία παραδοσιακά θεωρείται το κέντρο αν θέλετε, των μικρών κρατηδίων οπότε ε, πραγματικά ως Τουρκία εμείς ε, εκπροσωπούμε και συμβολίζουμε αν θέλετε ε, την, ακριβώς την υπεράσπιση των μικρών πόλεων εναντί των ευρύτερων δικαιωμάτων. αλλά εντάξει αυτό το λέω λίγο αστευόμενο τώρα έρχομαι στο διατάφτα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτή της ευλογικής περίοδου όπως ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι αν συγκρίνουμε τα πράγματα με το πώ είχαν πριν από πέντε χρόνια, διαπιστώνουμε ότι μετά από την χρηματοπιστωτική κρίση επιτύχαμε πολλά σε ό,τι αφορά τη σταθεροποίηση του τομέα και ακριβώ τη μείωση των ε, κινδύνων για την επιβάλληση των ε, φορολογούμενων πολιτών, έτσι ώστε να αναλάβουν την ευθύνη του οι ίδιε οι τράπεζε. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω και κάτι ακόμα ε, το οποίο δεν ακούστηκε σήμερα εδώ, αλλά αποτελεί τμήμα των συζητήσεων που κάνουμε κατά του τελευταίου μήνε. Ε, ε, και αυτό είναι το Brexit. Εσεί λοιπόν βλέπουμε να αναφέρεστε συχνά ότι δεν αποτελεί κάποιον εγγενή κίνδυνο αποσταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού μα συστήματο το Brexit. Ότι δηλαδή είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Μου αρέσει να το ακούω και με καθησυχάζει. Αλλά διερωτώ με, εμεί δηλαδή από την πλευρά τη πολιτική ε, ανησυχούμε υπερβολικά, γιατί ορισμένε περιπτώσει, ε, σε ορισμένε μάλλον περιπτώσει, ε, ή υπερβάλλουμε σε ό,τι αφορά τους κινδύνου που βλέπουμε ή ενδεχομένως εσείς να είστε ακριβώς πιο καθησυχαστικοί στα σχόλιά σας αλλά βλέπετε και εσείς σε σχόλια ε, αλλά από εκεί και μετά ε, να πω ότι πριν ε, από εβδομάδες ε, προβήκαμε σε κάποιους ε, διορισμούς ε, σε υψηλές θέσεις και διαπιστώσαμε εκεί ότι σε όλους αυτούς τους διορισμούς δεν υπήρχαν γυναίκες. Οπότε εσείς που είχατε αναλάβει τώρα τα χρέη προέδρου στο πλαίσιο της νέας περίοδου. Θα ήθελα να μας πείτε τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να έχουμε την ανάληψη περισσότερων θέσεων, υψηλότατων κορυφαίων θέσεων από την πλευρά των γυναικών έτσι ώστε δηλαδή να ε, ε, διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε μόνους, μόνο άνδρες οι οποίοι μπορούν να έχουν πολλά προσόντα, αλλά ε, χρειάζονται και γυναίκες. Πολλά λέμε για την Γερμανία. να επισκεφτείτε όλες αυτές τις περιοχές της Γερμανίας τις οποίες αναφερόμαστε εδώ. Λοιπόν, σχετικά με το Brexit, το σχόλιο μου και το προηγούμενο κάποιοι το πήραν εκτός πλαισίου. Εμένα με ρωτήσανε για την προετοιμασία του τραπεζικού κλάδου. Και νομίζω ότι ο τραπεζικός κλάδος, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος έχει προετοιμαστεί. Κάποιοι θα μπορούσαν να είχαν ε, προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα. Αλλά είναι και λογικό οι τράπεζες να περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τα θεσμικά όργανα σίγουρα ετοιμάστηκαν ε, τα διάφορα συμβούλια με διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους μηχανισμούς ε, εξυγίανσης. Έχουμε συνομιλήσει και με τους Βρετανούς ομολόγους μας. Το Brexit είναι θλιβερό και το Brexit θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Αλλά τον επικεντρωνόμαστε μόνο στο κατά πόσο κίνδυνος έρχεται για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή υπάρχει κίνδυνος για οικονομική κρίση γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι, εκεί το σχόλιο μου ήταν ότι έχουμε προετοιμαστεί αξιοπρεπώς και αν διαπιστώσουμε ότι λείπει κάποια άδεια για κάποιον, εγώ δεν θέλω να δω κανέναν να λέει ότι εγώ θα αφήσω το σύστημα να εκραγεί. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει ποια είναι η επίπτωση στην πραγματική οικονομία που στη συνέχεια επηρεάζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Και πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάντα πολύ καλή συνεργασία με τους Βρετανούς ομολόγους μας, την Τράπεζα της Αγγλίας, για παράδειγμα. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα συνεχιστεί, είτε μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι καλώς ποτέ δεν ήταν στην Τραπεζική Ένωση, είτε είναι εκτός Ευρώπης, όπως έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τους Αμερικανούς ομολόγους μας. Τώρα, το δεύτερο σχόλιο σας όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Εντάξει, ναι, προφανώς υπάρχει επιλογή, αλλά αυτό που κάνουμε είναι ότι κοιτάμε τη δικιά μας οργάνωση. Και έτσι έχω την ευκαιρία να ενθαρρύνω όλες τις γυναίκες με τα κατάλληλα προσόντα να είναι υποψήφιες για τις επόμενες θέσεις. Μόλις έχουμε δημοσιεύσει θέσεις για δύο μέλη του Συμβουλίου μας και ε, τον Αντιπρόεδρο, το οποίο θητεία λίγη στα τέλη της χρονιάς και έχω αρχίσει να το φωνάζω παντού όπου πηγαίνω και να λέω βάλτε υποψηφιότητα Εφόσον υπάρχουν γυναίκες που διαθέτουν τα προσόντα και το θέλουν παρακαλώ βάλτε υποψηφιότητα. Γιατί τελικά εμείς επιλέγουμε ανάμεσα στους υποψηφίους που έχουν υποβάλει την υποψηφιότητά τους. Αλλά βέβαια αυτό που σας λέω είναι ένα μικρό κομματάκι μόνο της όλης συζήτηση εννοείται. Για άλλη μια ερώτηση, ο κύριος Κέρχον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία ε, δεύτερη, ένα μάλλον δεύτερο ερώτημα σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλιση των ε, καταθέσεων, καθώς το αναφέρατε. αναφερθήκατε στη θέση του BMF, του δικού μας ταμείου δηλαδή και της γερμανικής κυβέρνησης, είναι ότι χρειάζεται ακριβώ το πλαίσιο του νέου πλαισίου να υπάρξει σε κρατικό, σε εθνικό επίπεδο ακριβώ αυτή η εξασφάλιση Εσεί είπατε ότι θα πρέπει ε, να προβούμε περαιτέρω στις προσπάθειες για την ολοκλήρωση τη χρηματοποιητική ενιαία αγορά, αλλά αν θέλουμε πράγματι να ακολουθήσουμε αυτά τα βήματα, τότε τίθεται το ερώτημα ε, του ε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε μέσα στο οποίο θα έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του έντις. Ελπίζω το έντις να αρχίσει να εφαρμόζεται σύντομα. Και το ελπίζω πραγματικά. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά όσον αφορά την εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων, αλλά τα εθνικά συστήματα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχει πρόβλημα μία τράπεζα, άρρητα υπάρχει ο κίνδυνος σε μια μικρή χώρα μέλος ή χώρα μέλος που φιλοξενεί την τράπεζα τι μπορεί να πει. Η δικιά μου αγορά κινδυνεύει, οπότε αποφασίστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τελικά η διάσωση. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη συζήτηση για τον επιμερισμό κινδύνου και την μείωση του κινδύνου. Μείωση κινδύνου και επιμερισμός κινδύνου. Αν περιμένετε να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο και πάντα σκέφτεσαι ότι μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο τελευταίο στάδιο, δεν ξεκινάτε ποτέ. Λοιπόν, ελπίζω να ξεκινήσει και να προχωρήσει η συζήτηση για το ΕΝΤΙΣ και στο Συμβούλιο, στην Ειδική Ομάδα Εργασίας, για να αποφασιστεί κάτι. Εδώ θα είναι για την επόμενη θητεία φαντάζομαι. Πάντως το έντις είναι ένα λογικό βήμα. Χρειάζεται, μπορείτε να κάνετε πολλά σε εθνικό επίπεδο και αυτό και εκείνο και το άλλο, αλλά το τραπεζικό πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Ο κύριε Μπερές. Ναι, αν μπορώ να πάρω ξανά το λόγο, ευχαριστώ. Κύριε Κένινγκ, ε, γιατί μου απαντήσατε στην πρώτη μου ερώτηση και προβληματίστηκα. Μου είπατε ότι η υπόθεση Δαρκάς ήταν το 2012, δεν είχαμε τους κατάλληλους μηχανισμούς στη διάθεσή μας κλπ. Αλλά εγώ δεν σας ρωτάω αυτό. Σας ρωτάω, η Μάλτα Δερκάς που είδαμε ότι ήταν η Γενική Διεύθυνση Κόμου που ασχολήθηκε η ερώτησή μου είναι εξή. Σε αντίστοιχη περίπτωση στο μέλλον, δεν νομίζετε ότι το Ταμείο Εξυγίανσης πρέπει να ασχοληθεί από την αρχή με την αξιολόγηση της κατάστασης και να δει τι γίνεται με την κινητοποίηση εθνικών πόρων από την εγγύηση καταθέσεων. Απάντηση. Όπως πάντα ρωτάτε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Εύκολα θα έλεγα ότι η τράπεζα αυτή ήταν μια μικρή τράπεζα. Υπό εθνική εποπτεία σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε σήμερα. Αλλά αυτό το οποίο βασικά θέλετε να ξέρετε είναι να πάμε τρία βήματα πιο πέρα, να δούμε τι γίνεται με την διαφοροποίηση στο πλαίσιό μας. Έχουμε την αρχή εξυγίανσης, που είναι το Συμβούλιο Εξυγένση, που έχει πρόσβαση στο Ταμείο Εξυγένση, αν χρειαστεί να εκτελεστεί απόφαση εξυγένση. και συγχρόνως έχουμε και εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων που ασχολούνται με την προστασία των ε, αποταμιευτών. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορές. Για την τάκα, είχαμε το ίδιο μέγεθος τράπεζας, τα ίδια στοιχεία σήμερα, θα ήταν εθνική η απόφαση βάσει του συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Υπάρχει βέβαια και μια ρήτρα που λέει ότι αν η Εθνική Αρχή αποφασίσει ότι δεν είναι θέμα εθνικό, αλλά είναι θέμα εξυγίανσης, έτσι, που έχει να κάνει ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι η τράπεζα, ε. τότε θα μπορούσαμε να πάμε για εξυγίανση και τότε εμείς θα αναλαμβάναμε και θα εμπλεκόταν και το Ταμείο Εξυγένσης, αλλά είναι αρκετά πιθανό. Αυτό δηλαδή βασικά που λέτε είναι ποια είναι η διάκριση ανάμεσα στα συστήματα αγγίσης καταθέσεων και τους μηχανισμούς εξυγίανσης. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο ήδη να εναρμόσουμε το έντις. Φανταστείτε τώρα να πούμε ότι το βάζουμε υπό ένα όργανο. Καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, και λέει η κυρία Κένινγκ, ε, για τα Χριστούγεννα ίσως. Εγώ δεν ε, πολύ πιστεύω, λέει η κυρία Μπερές, οπότε μην μου λέτε για τα Χριστούγεννα. Εγώ θέλω να ξέρω υπάρχει στρατηγική για την εξυγίανση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ξεκινάμε από τα εθνικά συστήματα. Μπαίνουμε σε μια λογική θα πληρώσει το κράτος ή όχι, που σημαίνει ότι τελικά δεν υπάρχει αναρμόνιση, δεν υπάρχουν ε, τα ίδια για όλους Οπότε λέτε εσείς ότι έχετε μια κατάλογο με επιθυμίες για το τι θέλετε να πετύχουμε στο μέλλον, αλλά εδώ υπάρχει κάτι πολύ βασικό. Η μη γενική διεύθυνση βασίζεται ε, στο κατά πόσο είναι ε, θέμα των κρατών ή όχι και μετά αποφασίζει για την εξήγηση ακόμα και αν νομικά δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα υπάρχει εδώ ένα θέμα σε αυτή τη διάκριση. Πώς γίνεται. Απάντηση. Να συμφωνήσω μαζί σας η ανακοίνωση της τράπεζας έχει να κάνει με το πώς θα εξετάσει το θέμα αυτό η Γενική Διεύθυνση και κατά πόσο όντως παρεμβαίνει η εξυγίανση ή τα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Συμφωνώ ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε περισσότερο, ναι. Συμφωνώ με αυτό. τελειώνει ο κατάλογος ε, καταναλωτών. Ο κύριος ε, θέλει τώρα το λόγο. Ο κύριος Τρεμόσα, εγώ έρχομαι από τη <laughs> Βαρκελόνη, ε, αλλά πάντως πριν από χίλια χρόνια η, χώρα μου, η πόλη μου ήδη συμμετείχε σε αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό project και ήταν συνδεδεμένη κατά κάποιο τρόπο με το ανώβερο. και ο Έρνστ Ιούγκερ μου είναι ιδιαίτερος προσφυλής ε, και στα 100 του χρόνια θυμάμαι ότι ο Χέλμουντ Κόρ και ο Φρανσουά Μιτεράν ε, πήγαν μαζί να του ευχηθούν χρόνια πολλά γιατί ε, ήταν ένα σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Συμβίωσης. Μια ερώτηση. Χτες είχαμε εδώ τον Λουίς Δεγκίντος από την NCB και τον ε, ε, ρωτήσαμε να μας πει κάποιες συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις γιατί όλοι μας ρωτάνε από τις πόλεις μας θα κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη τράπεζα, στους επιτηρητές κλπ νομίζω ότι θα πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό, γιατί δεν ακούμε συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εσείς μιλάτε για την ε, Banco Popular εκεί είχατε 10 ώρες για να αποφασίσετε ε, και φαίνεται ότι πολλά πράγματα μαγειρεύονται ήδη στις πρωτεύουσε και από ό,τι φαίνεται μονάχα 10 ώρες ε, έχετε για να συζητήσετε και μετά οι υπουργοί λένε ωραία, εγώ δεν έχω τίποτα να πω, πηγαίνετε στις Βρυξέλλες, πηγαίνετε στην Φραγκφούρτη και μετά κλείνει το θέμα. Βεβαίω καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να αποκαλύψετε τον τρόπο και να δώσετε πληροφορίε, αλλά κάπω πρέπει να βελτιωθεί αυτό. Όσον αφορά την Banco Popular, αν τώρα έφτανε σήμερα το θέμα αυτό σε εσά, θα κάνατε κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ. Να προσθέσω ότι υπάρχει και ένας ε, Ισπανός ε, συγγραφέας που ζει στην, ε, στο Ανόβερο και έχει γράψει το βιβλίο «Πάτρια», αλλά δεν θα πω το όνομά του γιατί δεν μπορώ να το προφέρω. Τι θα κάναμε κάτι διαφορετικό αν έφτανε σήμερα η υπόθεση της Banco Popular σε εμά. Όχι, δεν θα κάναμε κάτι διαφορετικό. Κάναμε ακριβώς αυτά που έπρεπε και ε, αυτά τα μαγειρέματα που λέτε. Ε, κοιτάξτε, η Φραγκφούρτη δεν είναι ούτε πρωτεύουσα χώρας ούτε πρωτεύουσα ομόσπονδου κρατηδίου, αλλά ε, οι Βρυξέλλες είναι η πρωτεύουσα του Βελγίου, είναι ε, η πρωτεύουσα της Ευρώπης και εκεί ελήφθη η απόφαση. Ευχαριστώ. Ο Σβάν επίση θέλει, Σβάν ε, αφού υπάρχει χρόνος, πράγμα πολύ σπάνιο, ε, γιατί είμαστε λίγοι τώρα, οι περισσότεροι έχουν πάει στις ε, χώρες τους. Δεν ξέρω, Ραμόνα, αν ξέρεις πόσο άσχημα αυτό κινήθηκε ε, και φέρθηκε ε, στην αρχή της δημοκρατίας ε, και στα πλαίσια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. εγώ τα ξέρω όλα αυτά και γι' αυτό πολύ προσεκτικά αντιμετωπίζω το θέμα. Εν πάση περιπτώσει όμως. Με ενδιαφέρει περισσότερο το MRL. Και ξεκινήσατε άλλωστε την παρέμβασή σας με αυτό. Είσαστε αρκετά επικριτικοί όσον αφορά κάποιες αλλαγές που συζητήθηκαν και εν τέλει συμφωνήθηκαν. Ενδιαφέρον θα ήταν να μας πείτε τώρα Ποια είναι η αξιολόγησή σας, δηλαδή είπατε ότι στο παρελθόν είπατε ότι οι νέοι κανόνες MRL και τα phishing option ε, θα μπορούσαν να οδηγήσει σε κατακαιρματισμό ε, ε, εξουσίας και ότι στην Ευρωζώνη θα είχαν μικρότερη δυνατότητα απόσβεσης κραδασμών οι τράπεζες. Τι έχετε να μας πείτε για αυτό. Το MRL εστιάζει βεβαίως σε μεγάλες και μεσαίες τράπεζες. Πώς βλέπετε όμως να, ε, με ποιο τρόπο βλέπετε να έχει επιπτώσεις στις μικρές τράπεζες. Απάντηξη. Όσον αφορά τη λεγόμενη phishing option, η άποψή μου δεν έχει αλλάξει. Θα πρέπει να δούμε όταν θα εφαρμόσουμε το νέο πλαίσιο εγώ είπα ότι θα πρέπει να ε, ε, επιτηρήσουμε την κατάσταση όταν θα ε, εφαρμοστεί το MRL και να δούμε πώς θα πάει. Το δεύτερο για τις μικρές τράπεζες. Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εάν χωρίσει κανείς ε, τις, ε, και καθορίσει τις τράπεζες, γιατί ήδη είναι δύσκολο να καθορίσει κανείς ποια είναι η μικρή τράπεζα, ότι ε, θα υπάρχει σταθερό MRL ίσως και στον πυλώνα 1. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα ή λιγότερα. Οι μεσαίες τράπεζες θα πάνε στο πυλώνα 2 και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Και όταν πια μιλά κανείς για τις πολύ μικρές μικρές ε, τράπεζες. Εκεί δεν υπάρχουν απαιτήσει MRL, γιατί για αυτές, αν κάτι δεν πάει καλά, τότε μπαίνουν στην αφαιρεγγιότητα και όχι στην εξυγίανση και επομένως δεν εμπίπτουν στο MRL που στην ουσία είναι κεφαλιακές απαιτήσεις. Βεβαίως θα πρέπει να παρακολουθούμε, να επιτηρούμε την κατάσταση και να δούμε και πώς το μεσαίο στρώμα των τραπεζών έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει το MRL γιατί διαφορετικά δεν, ε, ε, ούτως ή άλλως δεν έχει εναλλακτική Νομίζω ότι τώρα είμαστε ακόμα σε φάση επιτήρησης. Ε, πάντως ε, δεν έχει αλλάξει η θέση μου όσον αφορά τη λεγόμενη fishing option. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κιόνικ. Ε, ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτήν τη συνάντηση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί για μία ακόμα φορά δεν διστάσατε να έρθετε, να είστε στη διάθεσή μας. Με μεγάλη χαρά σας είχαμε εδώ ε, και να πούμε ότι έχουμε δουλέψει πολύ καλά από την αρχή του ε, μηχανισμού εξυγίασης. Αυτή είναι η τελευταία μου συνεδρίαση. Εδώ και 10 χρόνια δουλεύω στην Επιτροπή και συμμετέχω σε εργασία της Επιτροπής ΕΚΟΝ με πολύ δραστήριο τρόπο και πιστεύω και πρέπει να το πω ότι πολλή δουλειά έχει κάνει αυτή η Επιτροπή έτσι ώστε ε, να ε, είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πιο ασφαλή και να λειτουργούν σε ένα ασφαλέστερο και υγιέστερο πλαίσιο. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για την μεγάλη υποστήριξη γιατί δεν θα τα είχαμε καταφέρει αυτά χωρίς την κοινή προσπάθεια. Ευχαριστώ.

Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να περάσουμε στο σημείο 20. Στο σημείο 20 λοιπόν είναι ο διαρθρωμένος διάλογος με τον κύριο Νταμπρόφσκι που είναι ο αντιπρόεδρος για τον διάλογο για το ευρώ, οικονομική σταθερότητα, κεφαλαιακή ένωση κλπ. Καλώς ήρθατε και πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκι υπό την ιδιότητά του που είναι επίτροπος υπεύθυνος για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα φέτος. Επιτρέψτε μου λοιπόν εκ μέρους του Ισακό να τον συγχαρώ που, για ό,τι καταφέραμε, δηλαδή για την νομοθεσία αυτή που εγκρίθηκε και φρόντισε και ο πρόεδρος μας ο κ. Γκαλτιόρη γι' αυτό. Πάντως δεν θα καλύψει όλες τις πτυχές του χαρτοφυλακίου του, η ΕΚΟΝ προσπαθεί να βρει μια ημερομηνία για να έρθει και ως ε, πρόεδρος για τον κοινωνικό διάλογο στην Ευρωζώνη. Θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, 10 λεπτά πρώτα απ' όλα ο Επίτροπος για την εισαγωγή και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Υπάρχουν κάποια κενά, οπότε θα μπορέσουν οι πολιτικές ομάδες να ρωτήσουν ξανά και ξανά και μετά θα έχουμε και κάτι βέβαια. Παρακαλώ λοιπόν κύριε Ντομπρόφσκης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Πράγματι, όπως είπατε και εσείς, σήμερα είναι ο τελευταίος διαρθρωμένος διάλογος που έχουμε μαζί. Πριν λοιπόν αρχίσω, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μαζί τα τελευταία 4,5 χρόνια. Όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα, λοιπόν, πέρα από τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που εμπλέκονται, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των ε, πολιτών, διότι οι επιχειρήσεις επενδύουν, ε, απασχολούν εργαζόμενους. Χρειάζεται μια καλά διαρθρωμένη και οργανωμένη χρηματοπιστωτική αγορά. Επίσης, η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα καταφέρουμε να έχουμε σταθερά χρηματοπιστωτικά ή όχι. Έχουμε πετύχει πολλά μέχρι τώρα, χάρη και στην δικιά σας σκληρή δουλειά και δέσμευση. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πιο καθησυχασμένοι τώρα εν ώψη των επόμενων ευρωεκλογών. Ας αρχίσω με την κεφαλαϊκή αγορά. Από ε, τα, τους 13 τομείς που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 11 έχουν ήδη συμφωνηθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα επιτεύγματα αυτά είναι συγκεκριμένα βήματα για μια νέα αγορά κεφαλαίων που θα προσφέρει πραγματικά ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλω να συγχαρώ την ε, δικιά σας Οικονομική Επιτροπή για την πρόσφατη συμφωνία όσον αφορά την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών που είναι μια ε, σχετική πρόταση με τις κεφαλαικές αγορές και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεισηγητές την κυρία Μπερέση και τον κύριο Κάρας. Δεν φτάνει να έχουμε ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανονισμών. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις χώρες μέλη. Πρόκειται για μια πολιτική συμφωνία, η οποία είναι ένα σημαντικό βήμα για περισσότερη ε, ομοιομορφία και για βελτίωση των κανόνων όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την καταπολέμησή της δηλαδή. Θέλω ευχαριστώ επίσης την εισηγήτρια την κυρία Χούμπνερ για την πρόσφατη συμφωνία όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους και την εποπτεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και τον κύριο Λάγκεν για το Εμμύρ Ρεφίτ. Και επίσης την κυρία Σίνμπερνς και τον κύριο Βίντερς για την έκθεσή τους όσον αφορά ε, το CCP. Υπάρχουν βέβαια και άλλες προτάσεις όσον αφορά την ε, κεφαλαϊκή αγορά. Υπάρχει η έκθεση της κυρίας Σάντερ όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, από τον κύριο Καλφέτ Σαμπόν έχουμε και τη νέα προσέγγιση όσον αφορά την αφαιρεγγιότητα. Χάρη στη δουλειά επίσης του κύριου Φέρμπερ έχουμε ε, καταλήξει σε νέους κανόνες για τις επιχειρήσεις τις επενδυτικές και χάρη στην κυρία Σοφία Χετβέλτ συμφωνήσαμε και για ένα νέο πανευρωπαϊκό συνταξιδοτικό προϊόν. Συμφωνήσαμε επίσης να βελτιώσουμε και την ε, επενδυτική αγορά και σε αυτό βοήθησε ο συγκεκριτής ο κύριος Κλίντς. Και για τα καλυμμένα επίσης ομόλογα ο κύριος Μπέρντ Λιουκ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν προχωρήσει. Πρόκειται δηλαδή για συμφωνίες που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα για την τιτλοποίηση. Τέλος, θέλω να καλωσορίσω επίσης και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όσον αφορά το crowdfunding, τις διάφορες πλατφόρμες crowdfunding που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ενιαία διοδότηση με την βοήθεια των εισηγητών Fox και Νακτιγκέλ. Ελπίζω οι χώρες μέλη επίσης να αποφασίσουν σύντομα και να προχωρήσουμε επίσης για να προσφέρουμε και υπηρεσίες πληρωμών πιο φτηνές παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες μέσω του κανονισμού για τις διασυνοριακές πληρωμές. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό την εισηγήτρια την κυρία Εύα Μέιντελ. Όταν ξεκινήσαμε τη δουλειά μας για τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά, λίγοι πίστευαν ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και όμως με τις προσπάθειες των εισηγητών, του κ. Πολ Τάν και της Νίνα Τζιλ, Πρόσφατα καταλήξαμε σε συμφωνία για δύο από τις τρεις προτάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Η πρώτη έχει να κάνει με την διαχείριση των επενδύσεων και πώς θα λαμβάνονται υπόψη το θέμα της βιωσιμότητας της επενδύσεις και το δεύτερο έχει να κάνει με τις προδιαγραφές υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Όσον αφορά την πρότασή μας λοιπόν για την ε, ταξινόμηση των ε, ε, χρηματοπιστωτικών παραγόντων που είναι βιώσιμοι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην ε, Ολομέλεια την ε, προηγούμενη εβδομάδα και ευχαριστώ για αυτό τους συζητητές ΕΚΑΟΤΟ και τι Κάινεν. Έρχομαι τώρα στην Τραπεζική Ένωση. Έχουμε προχωρήσει πολύ για να περιορίσουμε τους κινδύνους και να ενισχύσουμε την αντοχή του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Κλάδου. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε πετύχαμε πολιτική συμφωνία για το τραπεζικό πακέτο μετά από πολλού μήνε δύσκολων διαπραγματεύσεων. Οπότε ευχαριστώ πολύ του ηγητέ Χόκμαρ και Σίμων για το έργο τους όσον αφορά αυτό το πολύ σημαντικό πακέτο για τη μείωση κινδύνου. Μαζί επίσης προχωρήσαμε πολύ και όσον αφορά τα μη ξεπηρετούμενα δάνεια. Το μέσο επίπεδο των μη ξεπηρετούμενων δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα είναι στο 3,3% το, τέταρτο, το τρίτο τέταρτο δηλαδή του 2018. Επίσης είχαμε συμφωνία τον Δεκέμβριο για τον μηχανισμό προστασίας των προληπτικό όσον αφορά τα μη ξεπηρετούμενα δάνεια και αυτό χάρη στους ηγητές την κυρία Λάγκια και τον κύριο Γκουαλτιέρη. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως ε, τη δουλειά μας, γι' αυτό και χαίρομαι πολύ και σας ενθαρρύνω στις προσπάθειές της για να προχωρήσουμε περισσότερο όσον αφορά τις δευτερογενείς αγοράς για τα μη ξεπηρετούμενα δάνεια. Ελπίζω να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην επόμενη θητεία. Και σας ευχαριστώ πολύ επίσης και για ό,τι κάνατε για τα κρατικά ομόλογα και την τιτλοποίηση χάρη στον εισηγητή τον κύριο Γιώνας Φερνάντες. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει βοηθήσει πάρα πολύ για την ε, διαφοροποίηση όσον αφορά το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών με σταδιακό τρόπο σιγά σιγά. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, ευχαριστούμε πολύ για τη συμφωνία. Όσον αφορά τον κοινό μηχανισμό προστασίας για, για το ενιαίο Ταμείο Εξυγένσης που εφαρμόζεται. Και επίση υπάρχει πρόσκληση όσον αφορά το έντυπο. Κυρίε και κύριοι, χρειάζεται περισσότερη δουλειά όμω. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Brexit που αποτελεί μια πρόκληση για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κλάδο. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή ενιαία. Επίσης, πρέπει να αναπτύξουν περισσότερο τις ευρωπαϊκές αγορές, ενισχύοντας την ικανότητά μας όσον αφορά τις πηγές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, τις υποδομές των αγορών και την εποπτεία των αγορών. Ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε περισσότερο και με την επόμενη Κομισιόν. Έπειτα, όσον αφορά το τραπεζικό κλάδο, βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από 10 χρόνια, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθειές μας για να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση έχουμε αρχίσει μια αξιολόγηση αντικτύπου ήδη όσον αφορά την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Βασιλεία 3. Έπειτα υπάρχουν νέες τάσεις όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια που επιταχύνονται και η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να έχει μια ισχυρή φωνή στην παγκόσμια σκηνή, γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε και το διεθνή ρόλο του ευρώ. Πρέπει να προσαρμόσουμε τις ρυθμίσεις μας βάσει των εξελίξεων στην τεχνολογία ε, και οι εξελίξεις αυτές μόλις αρχίζουν. Γι' αυτό λοιπόν περιμένω ότι θα γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα και πρέπει επίσης να ευθυγραμμίσουμε και τις χρηματοπιστωτικές ροές βάσει του στόχου μας που είναι μια οικονομία η οποία δεν καταστρέφει το κλίμα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ αρνητικές για μας αλλιώς. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Συγχαρητήρια και πάλι για το κοινό μας έργο για ό,τι πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και να ακούσω τα σχολιά σας. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν ξεπεράσατε καθόλου το χρόνο σας. Εξαιρετικό και όχι πολύ ε, σύνηθες. Ε, λοιπόν, ερωτήσεις και απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, Μάρκος Φέμπρε από, τους, ε, ε, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, εξ ονόματος ε, του ΕΛΚΕ θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω κύριε Αντιπρόεδρε για την εξαιρετική συνεργασία ε, που είχαμε στην προηγούμενη θητεία που τώρα τελειώνει. Ε, είχατε πραγματικά πολύ σημαντικές αρμοδιότητες ε, και ε, είχατε και τους φακέλους τους οποίους κληρονομήσατε κατά κάποιο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για όλα όσα κάνατε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, κάποιες ερωτήσεις θέλω να υποβάλω. Πρώτα απ' όλα, ε, όσον, αφορά, όσον αφορά τα πρίψ, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί και ε, λάβατε και ε, επιστολή από τρεις ε, οργανισμούς επιτήρησης για το θέμα αυτό και φαίνεται, φαίνεται ότι σε επίπεδο λιανικής υπάρχουν προβληματισμοί όσον αφορά τις απαιτήσει και τις προϋποθέσεις που πρέπει να γίνουν σεβαστές και για κάποια προϊόντα αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα όσον αφορά την κεφαλή αγορά. Θα πρέπει να ρυθμιστούν λοιπόν τα σημεία αυτά. Ε, δεύτερον, και επανερχόμαστε δυστυχώς ε, στη, στο Brexit. Η ΕΣΜΑ λέει ότι εάν το Brexit είναι σκληρό, τότε τουλάχιστον βράχει πρόθεσμα ε, θα υπάρξουν προβλήματα όσον αφορά ε, τις, ε, τα επιτόκια και όσον αφορά τους βασίλους κεφαλαίου και τα λοιπά. Μέχρι, ποια είναι η περίοδος επαναστόχευσης κατά τη δική σας άποψη, πόσος χρόνος θα χρειαστεί έτσι ώστε να ξεπερασούν τα προβλήματα. Ε, και άλλωστε ε, οι επιπτώσεις μπορεί να ε, διευρυνθούν και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά τον πιθανό αντίκτυπο και τι μπορούμε να κάνουμε. Κυρία Αντιπρόεδρε, θέλετε να απαντήσετε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτη ερώτηση σε σχέση με τα corporate bonds, αυτά τα PRIPS που λέμε. Ξέρετε ότι η διαφάνεια των επενδύσεων ε, ε, λιανικής ε, υπάρχει και ότι υπόκεινται όλα αυτά τα προϊόντα στους κανόνες της κεφαλαίου αγοράς κλπ. Η αξιολόγηση σε περίπτωση ε, που η επένδυση ε, υπόκειται στα πρίψ, ε, πρέπει να γίνεται αναπερίπτωση. Στην ουσία δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει το όνομα, δεν είναι δυνατόν να γίνει εξάντε και με ασαφή τρόπο ο υπολογισμός το ίδιο ισχύει ε, και για τα corporate bonds. Κάποια από αυτά τα ομόλογα μπορεί να εμπίπτουν στα μπρίψα, αλλά εταιρικά ε, ομόλογα να μην εμπίπτουν και να αφορούν συγκεκριμένες συμβατικές ε, συμφωνίες. Αυτό που καθορίζει ο κανονισμός ε, είναι ότι θεωρεί τις επενδύσεις λιανικής ε, σαν επένδυση της οποίας η επιστροφή υπόκειται στην διακύμανση. Δηλαδή το ποσό το οποίο ε, θα πληρωθεί εν τέλει στον επενδυτή δεν είναι σαφές από την αρχή. Απ' την άλλη πλευρά μας ενδιαφέρει βεβαίως και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ε, την ε, συνεκτική αντιμετώπιση όλων αυτών των προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των εταιρικών ομολόγων. έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, αθέλητες επιπτώσεις. Όσον αφορά τώρα την δεύτερη ερώτησή σας, όσον αφορά το Brexit. Για το Brexit, να πω το εξής. Ξέρουμε ότι υπάρχει ε, κίνδυνος την 12η Απριλίου το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, συμφωνία. Ο κίνδυνος ε, υπάρχει, είναι υπαρκτός και στην Κομισιόν έχουμε ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια αποχώρηση no deal, χωρίς συμφωνία υπάρχουν κάποιες ε, ε, περιπτώσεις όπου ο συστημικός κίνδυνος ε, για πρόκληση χρηματοπιστωτικής αστάθειας είναι μεγαλύτερος και κατά αυτήν την έννοια ενδεχομένως θα ληφθούν κάποια κάποια πρόσκαιρα μέτρα. Αλλά φυσικά δεν θα είμαστε ε, σε θέση και δεν θα έχουμε την δυνατότητα να μετριάσουμε οποιοδήποτε είδους ε, οικονομική ε, ζημία. Οπωσδήποτε θα υπάρξουν προβλήματα, disruptions αλλά οπωσδήποτε σιγά σιγά οι αγορές θα προσαρμοστούν στην νέα κατάσταση και άλλωστε και οι αγορές προετοιμάζονται εδώ και αρκετά χρόνια ξέρουν ότι έπρεπε να προετοιμαστούν για διάφορα ενδεχόμενα και διάφορα σενάρια μεταξύ των οποίων και αυτό του Brexit υπάρχει και βεβαίως ε, εμείς για, οποιαδήποτε, για οποιοδήποτε ενδεχόμενο ε, συμβουλεύουμε όλους τους εμπλεκόμενους να προετοιμαστούν ε, κατάλληλα. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια σε τελική κινδύνη που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε θεσμικό επίπεδο και με αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων, σε επίπεδο, σε επίπεδο κρατών μελών. Όσο δε αφορά τα ζητήματα της ε, ΕΣΜΑ, και την ανταλλαγή πληροφοριών και την ε, ε, διαφάνεια των απαιτήσεων να σας πω ότι ε, επ' αυτού εργάζεται η ΕΣΜΑ και έχει δώσει και κάποιες αποσαφηνήσεις σε σχετικές ανακοινώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και βεβαίως όλοι είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να συνεργαστούμε με την ΕΣΜΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ε, για αυτή την απάντηση για τους σοσιαλιστές τη Μπερές. Κύριε Αντιπρόεδρο, εξ ονόματος ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια ολόκληρη θητεία συνεργασίας, θητεία κατά τη διάρκεια της οποίας οι αρμοδιότητές σας διευρύνθηκαν ε, και οπωσδήποτε όλοι, συν, ε, όλοι μαζί προσθέσαμε κάποια στοιχεία στο νομοθετικό οπλοστάσιο. Αναθεώρηση λοιπόν των εποπτικών αρχών και εδώ το αναφέρατε αυτό ε, και σας παραπέμπει στην αρχή της θητείας όπου γινόταν οι πρώτες συζητήσεις για την κεφάλαια αγορά και εγώ σας έλεγα ότι χωρίς επιτήρηση ε, ε, δεν μπορεί να υπάρξει η δημιουργία κεφαλαίου αγορών. Αντιμετωπίσατε αντίσταση υπερβολική μερικές φορές από τα κράτη-μέλη. Ερώτηση όμως. Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτοί που θα μας διαδεχθούν και θα σας διαδεχθούν θα έχουν την διάθεση, τη θέληση να ξανανοίξουν το θέμα ε, της επιτήρησης. Αλλά να σας δώσω δύο παραδείγματα το ζήτημα του εσωτερικού μοντέλου ε, στις ασφάλειες. Όλοι ξέρουν και όλοι γνωρίζουν ότι ε, το EIS, το αντίστοιχο της Επιτροπής της Βασιλείας, ε, ε, εξετάζει από πολύ κοντά αυτό το θέμα του εσωτερικού μοντέλου. Τα κράτη-μέλη λένε, ας πούμε, ότι το εσωτερικό μοντέλο επιτηρείται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο, αλλά δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να πιστεύει ότι κάτι τέτοιο είναι αξιόπιστο. Πώς είναι δυνατόν να ξεπεραστεί λοιπόν αυτό το ε, ε, πρόβλημα, αυτό το εμπόδιο, εκτός και αν περιμένουμε την επόμενη κρίση για να γίνει αυτό υποχρεωτικό. Δεύτερο, η ερώτηση της ε, συνέχειας που δυστυχώς θα υπάρξει στο ενδεχόμενο Brexit. Ναι, μπορούμε να προωθήσουμε την επιτήρηση των CCP τρίτων χωρών, αλλά τι γίνεται με την επιτήρηση των CCP στο εσωτερικό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μερικές ε, χώρες μπλοκάρουν πλήρως την κατάσταση ε, και μας λένε να, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για την μετατόπιση αυτών των αντισταθμιστικών. Άρα τι θα κάνουμε εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματικά μια, μια ουσιαστική πραγματική κεφαλαία αγορά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εγώ έχω βαρεθεί πια να ακούω συνέχεια να αναμασούν οι Ευρωπαίοι ότι είμαστε υπέρ τη κεφαλαία αγορά και είμαστε υπέρ τη ένωση ε, των κεφαλαίων κτλ. Ναι, αλλά όταν πρέπει να βάλει κανεί το χέρι για να ανακατέψει το γλυκό, κανένα δεν βρίσκεται. Uh, <coughs> uh, okay. Uh, thank you for this question. Σας ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση, ήδη το έδειξα στις προκαταρκτικές, ε, στην προκαταρκτική στα προκατακτικά σχόλια που έκανα και σας είπα ότι από την πλευρά της Επιτροπής θέλουμε να έχουμε μια ή θέλαμε να έχουμε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση, ωστόσο τελικά το ε, τελικό αποτέλεσμα ήταν αποτέλεσμα πολιτικού συμβιβασμού. Σίγουρα πάντως πρόκειται για ένα χρήσιμο βήμα προς τα μπροστά, το οποίο δίνει στις σας ε, περισσότερες αρμοδιότητες και καλύπτει νέες περιοχές όπως ε, fintech, ε, δηλαδή βιώσιμη χρηματοπιστωτική, βιώσιμο χρηματοπιστωτικό κλάδο, η δραστηριότητα, sustainable finance, τα, τα CCP από τρίτους, τους κεντρικούς δηλαδή από τρίτες χώρες και ούτω καθεξής και ειδικότερα σε ό,τι αφορά του κεντρικού αντισυμβαλόμενου. Γνωρίζετε καλά τι συζητήσει που έχουν γίνει. Πάντω, ε, αν ε, ρίξουμε μια ματιά ε, πριν από μερικέ εβδομάδε, ένα-ενάμιση μήνα πριν, θα διαπιστώσουμε ότι μέχρι τόσο πρόσφατα δεν ήταν σίγουρο ότι θα καταφέραμε ε, τόση πρόοδο. Και γνωρίζατε που το Συμβούλιο που βρισκόταν κοντά στο να κάνει αυτό το διαχωρισμό δηλαδή του κομματιού της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε, και τελικά γνωρίζετε ότι εμείς αγωνιστήκατε από πλευρά της Επιτροπής αυτό να παραμείνει ένα ενιαίο πακέτο και να μην υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Σίγουρα δεν φτάσαμε εκεί που θέλαμε για μας για την Επιτροπή, αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα χρήσιμο πρώτο βήμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την επόμενη θητεία, και την επόμενη επιτροπή. Εγώ δεν μπορώ να προδικάσω βέβαια τι επιλογέ που θα, κάνω, αλλά, που θα κάνει, αλλά θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες της νέα επιτροπή προς την, ένωση των, την, την κοινή αγορά των κεφαλαίων γιατί ε, πρόκειται για κάτι το οποίο χρειαζόμαστε και το οποίο είναι απαραίτητο για την ευρωπαϊκή οικονομία γιατί παίζουν ακριβώς οι κεφαλαίων πολύ σημαντικό ε, ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες εδώ προς αυτήν την ενιαία αγορά κινούμενη σε διάφορους άξονες εδώ συμπεριλαμβανομένου ακριβώς και του, του, κομματιού της εποπτείας. Και θα ξεκινήσουμε προφανώς και τις εργασίες μας ό,τι αφορά το SS Review, αλλά σίγουρα αυτό πλέον θα αποτελέσει αρμοδιότητα της επόμενης επιτροπής να το κάνει. Δεν υπάρχει ομιλητή για λογαριασμό του ΙΣΕΡ. Για την άλλη, λοιπόν, ο κύριο Σάμονσον Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Ντομπροφστή, ε, για την πολύ καλή συνεργασία που κάναμε. Ήταν πραγματικά εύκολο το να βρισκόμαστε επαφή μαζί σα και σα ευχαριστώ για τη συνεργασία μα. Ε, πραγματικά καταφέραμε να καταλήξουμε σε μία σειρά από νομοθετικού ε, φατέλου και θα πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό το επιτευγμα. τώρα, έχω να θέσω κάποια ερωτήματα. Είδαμε ε, πω ο πρόεδρο Γιούγκερ αναφέρεται στην Ιταλική οικονομική ανάπτυξη, αλλά νομίζω πω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι η Ιταλία είναι η χώρα που επέτυχε το υψηλότερο ε, πρωτογενές πλεονάσμα τα τελευταία χρόνια. Ενώ ε, στην Ισπανία, για παράδειγμα, έχουμε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αλλά με βάση τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν, το πάνω από ένα τρίτο αυτής της οικονομικής ανάκαμψης, η αύξησης, οφείλεται στην αύξηση της δημόσιας δαπάνης. Και υπάρχει ε, και βέβαια το έτοιμα του 3% του ΑΕΠ. Οπότε βλέπουμε και αυτή την οικονομική κρίση ε, η οποία ενδεχομένω ε, να επέλθει για την Ισπανία ακριβώ γιατί γίνεται τόσο μεγάλη δαπάνη από τα δημοσιοοικονομικά πράγμα το οποίο μπορεί να ισχύσει ε, και αντίστοιχα και για την Ιταλία. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω αν ε, παρακολουθείτε αυτή την κατάσταση. Πάντω αυτό ε, με φέρνει στο να σχολιάσω την κατάσταση που ισχύει στα διαφορετικά κράτη-μέλη και ο κύριο Δεκίνητο, ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανέφερε χθε στην ομιλία του εδώ σε αυτή την επιτροπή ότι υπάρχει περιβολική προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών, πολλέ τράπεζε στην Ευρώπη Ωστόσο υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη στα οποία υπάρχουν μόνο δύο, τρει, 4 μεγάλε τράπεζε ενώ οι υπόλοιπε μικρέ τράπεζε έχουν εξαλειφθεί. Άρα λοιπόν ε, υπάρχει και ο κίνδυνο να, να οδηγηθούμε σε υπερβολική συγκέντρωση ε, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα επιτόκια τα οποία, και το πώ θα μπορούσαν να διαμορφωθούν σε ό,τι αφορά τη χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θα ήθελα να μου πείτε τι νομίζετε εσεί. Ε, Ευχαριστώ. για την πρώτη ερώτηση που είναι δευτερογενός του χαρτοφυλακίου μου. Πράγματι, αν κοιτάξουμε τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται. Διότι τα στοιχεία τα οποία εξακολουθούν να μας έρχονται μετά τις χειμερινές προβλέψεις φαίνεται ότι συνεχίζεται η επιβράδυνση και στις ε, προβλέψεις της άνοιξης ε, θα προβλέπεται χαμηλότερη ακόμα ανάπτυξη. Και αυτό έχει να κάνει με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, ε, κυρίως την Ιταλία θα έλεγα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Σε όλες αυτές τις χώρες δηλαδή υπάρχει χαμηλότερη ανάπτυξη. Είναι πολύ βασικό ως παράγον. Και κάτι άλλο το οποίο τονίζαμε πάντα με τις χώρες μέλη όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν τους καλούς καιρούς. Για τώρα είμαστε στο 7ο έτος ανάπτυξης, οπότε να φροντίζουν να εξοπλίζονται τώρα στους καλούς καιρούς των παχαίων αγελάδων για να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολους καιρούς. Η κατάσταση δεν είναι βέβαια ε, η ιδανική. Κάποιες χώρες μάλιστα βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση δημοσιονομικά και τους λέμε να χρησιμοποιήσουν τις, ε, τη δημοσιονομική τους πολιτική για να βελτιώσουν την κατάσταση χώρες που έχουν πολύ ψηλά ελλείμματα και χρέος, που φυσικά δυσκολεύονται να τα μειώσουν. Αλλά και αυτός είναι παράγοντας κινδύνου, όπως λέτε κι εσείς. Το παρακολουθούμε από κοντά. Για την άλλη σας ερώτηση όσον αφορά την συγκέντρωση των τραπεζών. Όπως γνωρίζετε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προκαταλαμβάνουμε εμείς, δεν λέμε πόσες τράπεζες πρέπει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι η αγορά και σε ένα βαθμό και χώρες μέλη που το αποφασίζουν αυτό. Όμως πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται διαφοροποίηση στον κλάδο των τραπεζών και μεγάλες ε, και λιγότερο μεγάλες και μικρές που να επικεντρώνονται στις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εμείς ακριβώς προσπαθήσαμε να εισάγουμε περισσότερη αναλογικότητα στο χρηματοπιστωτικό μας ε, τομέα και στις κανόνες ρύθμισης των ε, τραπεζών, ώστε να ρυθμίζονται οι τράπεζες αναλογικά με τους κινδύνους που ελοχεύουν. Και πιστεύουμε ότι αυτή η αναλογικότητα βοηθάει και δείχνει ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή την διαφοροποίηση στον κλάδο των τραπεζών στην Ευρώπη. Βέβαια χρειάζονται και ρήτρε ασφάλεια. Έχουμε έλεγχο συγχωνεύσεων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κάποια τράπεζα γίνει υπερβολικά ε, μεγάλη. Και επίση έχουμε υπόψη μα ότι πρόκειται για μια κίνηση, είναι κάτι ρευστό. Εξαρτάται από τον ανταγωνισμό, γι' αυτό και θέλουμε την Κεφαλαιακή Ένωση και το Φίνεξ ο τραπεζικός κλάδος θα συνεχίσει και ο ανταγωνισμός θα διατηρηθεί στον κλάδο. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο Σβέν Γκίγκολτ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπη, ήσασταν στην πρώτη γραμμή όταν αναλάβατε τη θέση σας για βιώσιμα βιώσιμους, χρηματοπιστωτικέ χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Όμως θα ήθελα να γνωρίζω τα εξή δύο. Πρώτον, όσον αφορά την οικολογική σήμανση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ήτανε μια δικιά σας φιλοδοξία αυτή. Και το ανακοινώσατε και πάλι τον Ιανουάριο σε μια ομιλία σας. Ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων σήμερα, πότε θα έχουμε την επέκταση αυτής της ε, οικολογικής σήμανσης και στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Δεύτερον, όσον αφορά τις εξελίξεις για τις προδιαγραφές των οικολογικών ομολόγων. Ε, υπήρξε μια πρόταση, αλλά τελικά καταλήγουμε σε status quo δεν είναι υποχρεωτικοί οι κανόνες, δηλαδή είναι πιο αδύναμοι ακόμα και από αυτούς που έχει υιοθετήσει η αγορά μερικές φορές. Η Κίνα, η Ινδία λέμε ότι θέλουμε να έχουν ε, υποχρεωτικές τέτοιες ρυθμίσεις και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς δεν θα πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή, δεν θα πρέπει εμείς να βάζουμε τις προδιαγραφές. Τώρα η τεχνική ομάδα εργασίας προτείνει μη δεσμευτικούς κανόνες. Τι περιμένουμε, το greenwashing να μας αναγκάσει να ρυθμίσουμε και να είναι άλλες χώρες του κόσμου στην πρώτη γραμμή γι' αυτό. Εμείς όταν πρόκειται για πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Οπότε θα κάνετε κάποια σχετική πρόταση για τη, στα πλαίσια της ε, κατεξοδότηση ρύθμισης. Απάντηση. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Αρχίζουμε με την πρώτη σας ερώτηση για την οικολογική σήμανση. Πράγματι, Το συμπεριλάβαμε αυτό στο πρόγραμμα δράση μας για τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και δουλεύουμε πάνω σε μια τέτοια οικολογική σήμανση για τους μικρούς επενδυτές. Ήδη έχει ξεκινήσει η δουλειά και σύμφωνα με το σημερινό χρονοδιάγραμμα η έγκριση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση είναι για τον Νοέμβριο του 2020 για την πρώτη κατηγορία προϊόντων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Και αυτή η πρώτη ομάδα θα έχει τα επενδυτικά ταμεία ε, και επενδυτικά προϊόντα, γιατί είναι αυτά ε, τα οποία κυκλοφορούν περισσότερο στην αγορά και μετά θα προβλέψουμε και άλλα προϊόντα σε ένα δεύτερο στάδιο. Αυτά σύμφωνα με τα σχέδιά μας. Έτσι, δεν θέλω να προκαταλάβω εδώ ότι θα κάνει η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι. Πάντως, η δουλειά συνεχίζεται και η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη θα βρει ότι η δουλειά έχει προχωρήσει πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά τις προδιαγραφές για πράσινο ομόλογα. Πράγματι, η τεχνική ομάδα πραγματογνωμοσύνης έχει ήδη παρουσιάσει την πρώτη της έκθεσή της και ζητάμε feedback τώρα. Και μάλιστα η προθεσμία λίγη αύριο. Βάσει αυτού του feedback λοιπόν και της τελικής έκθεσης της ομάδας αυτής της τεχνικής που αναμένεται για τον Ιούνιο θα δούμε ποιες είναι οι συστάσεις και θα σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα. Ίσως η αξιολόγησή μας να μην είναι τόσο επικριτική Σύμφωνα με την προσέγγιση της τεχνικής ομάδας, οι δικές μας προδιαγραφές πρέπει να βασιστούν στις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα πράσινα ομόλογα και την πρωτοβουλία για τα ομόλογα κλίματος. Η ομάδα αυτή πάντως βάζει τις προδιαγραφές με επαλήθευση, με ένα σύστημα πιστοποίησης για να ενισχυθεί η αξιοπιστία και να αποφεύγεται το greenwashing. Θα υπάρξουν και κίνητρα κατά πάσα πιθανότητα υπέρ των, ε, της έκδοσης πράσινων ομολόγων. Και σίγουρα υπάρχει και το θέμα της ταξινόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το οποίο νομίζω ότι ήμουν σαφής. Μετά, όσον αφορά τις κατεξοδότηση πράξης. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα δεν σχεδιάζουμε ε, κατεξοδότηση πράξης για τα πράσινα ομόλογα. Μπορούμε να το συζητήσουμε περισσότερο σε λεπτομέρειες και να δούμε πού μπορεί να χρειάζονται ακριβώς. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως θα αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα μετά την τελική έκθεση της ομάδας της τεχνικής που όπως σας είπα περιμένουμε τον Ιούνιο. Και τότε θα δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Θα δούμε δηλαδή αν τελικά χρειάζεται κάποια ή όχι. Ευχαριστούμε. Γκουέ δεν είναι εδώ. Μάρκο FDD τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις ε, για τον ε, ε, κύριο Ντομπρόφσκης. Πρώτα απ' όλα, μείωση κινδύνων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Ξέρουμε ότι επικεντρωθήκαμε κυρίως στον πιστοτικό κίνδυνο και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να ρωτήσω αν η Κομισιόν αξιολογεί επίσης και κάποια στοιχεία του, του κινδύνου που δεν έχουν ληφθεί αρκετά υπόψη. Έχουμε βεβαίως τις εποπτικές αρχές και την Κεντρική Τράπεζα που ε, αρχίζουν να λαμβάνουν υπόψη του τίτλους ε, δευτέρου ε, και τρίτου επίπεδου, κυρίως τα, τα παράγωγα τα οποία έχουν ε, ε, εμφανιστεί σε κάποιες ε, τράπεζες και με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά περισσότερο την Ιταλία. Θα ήθελα την άποψή σας όσον αφορά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ακύρωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε απαγορεύσει την ε, χρήση ε, της διατραπεζικής ε, διευκόλυνσης σε περίπτωση κατά την οποία έμπαινε σε κρίσιμη κατάσταση τράπεζα Τέρκας. Βεβαίως ακολούθησαν και μία σειρά γεγονότων που δημιούργησαν μεγάλη ζημία στο, στο ιταλικό σύστημα αύξηση των spread καθώς επίσης και την επίπτωση τύπου ντόμινο ε, για τράπεζες ε, όπως το Βένετο, η Μοντεπάσκι και τα λοιπά ε, και μεγάλες ζημίες δεκάδων δις στην Ιταλία και είναι πολλοί στην Ιταλία πλέον οι οποίοι θέλουν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένες εξηγήσεις. Ευχαριστώ. Απάντηση. Όσον αφορά την ε, πρώτη ερώτηση, μείωση πιστοτικού κινδύνου ε, στον τραπεζικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γι' αυτό μπορώ να πω ότι επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας σε όλα τα στοιχεία των τραπεζών, banking books, trading books. Είναι μεγάλη προτεραιότητα για μας αυτό. όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το είπα άλλωστε και στην εισαγωγική μου παρουσίαση. Έχουμε προχωρήσει στη μείωση, ικανοποιητικά στη μείωση των μη ε, ε, εξυπηρετούμενων ε, δανείων. Φυσικά η κατανομή αυτών των δανείων δεν είναι καθόλου ισομερής στα κράτη-μέλη και έχουμε ε, ακόμα αρκετές χώρες στις οποίες, ε, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο επίπεδο. Ναι, 40% στην Ελλάδα, 30% ε, περίπου στην Κύπρο είναι αυτές οι δύο χώρες οι οποίες ε, βρίσκονται πολύ πολύ μακρύτερα από τις άλλες όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ε, όσον αφορά ε, συγκεκριμένα την κατάσταση στην Ιταλία και η Ιταλία μείωσε το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων και μάλιστα με πολύ σημαντικό τρόπο τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν συζητούσε συγκεκριμένες διατάξεις. Τα τελευταία στοιχεία για το τρίτο τετράμινο του, του 2018 ε, η Ιταλία βρίσκεται στο 9,5% αντί του 12,5% ένα χρόνο πριν και για την Κύπρο επίσης έχουμε ε, ε, ε, τώρα 22% το 2018 ενώ ήταν πάνω από 30% το 2017 21,8 32,1. Όσον αφορά την άλλη ερώτηση για την απόφαση Τέρκας, το δικαστήριο αποφάσισε βάσει των στοιχείων της Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή εμείς μελετούμε ε, την απόφαση και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της. Ταυτόχρονα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε προγράμματα ε, ε εγγύησης καταθέσεων όπως αυτό το φόντο Ιντερμακάριο στην ε, Ιταλία σε, με την προϋπόθεση μόνο να μην ε, αποτελούν κρατική επιδότηση, πράγμα που συνέβη στην περίπτωση της τράπεζας ε, Τέρκας. Όσον αφορά τις μικρές ε, τράπεζες Ετρούρια, Μάρσετ, Γαρίφε και Ριτσέτε, Αυτές οι τράπεζες μπήκαν σε εξυγίανση το 2015 μετά από απόφαση της τράπεζας της ε, Ιταλίας. Ε, βεβαίως υπήρξε προστασία των καταθετών ε, και οι Ιταλικές αρχές συνεργάστηκαν επικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να λυθούν και προβλήματα τα οποία είχαν ε, σχέση με προβληματικές πωλήσει ομολόγων κλπ. Ε, ε, επίσης, πολύ καλή συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές όσον αφορά νέες προτάσεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι η σειρά μου να υποβάλω ερωτήσεις. Αναφερόμαστε σε μια σειρά από επιτεύγματα στον τομέα της οικονομικής σταθερότητας και της εποπτείας, αλλά βέβαια πρόκειται για επιτεύγματα τα οποία δεν έχουμε ολοκληρώσει. Πάντως θα ήθελα να αναφερθώ και σε περαιτέρω ζήτημα της δικής σα δηλαδή εδώ στο ξέπνομα του βρώμικου χρήματος. Ειδικότερα για παράδειγμα τα ζητήματα εκείνα της Danske Bank, ε, ε, περίπτωση του Αζερβαϊτζάν και ούτω καθεξής. Οπότε σας ερωτώ, δεν σας ανησυχούν αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις ε, στην οικονομική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, καθώς εσείς κατάγεστε και από μια χώρα της ε, Βαλτικής ε, θα σας ρωτήσω πώς μπορούμε να επιτύχουμε εδώ σημαντικές βελτιώσεις. Ένα δεύτερο ερώτημα ε, δεν μπορούν να είναι οι τράπεζοί μας καλύτερες από το, το, το σύνολο της οικονομίας μας και βλέπουμε λοιπόν ότι η οικονομική μας ανάπτυξη μετριάζεται λίγο και το Brexit θα επιφέρει ένα περαιτέρω πλήγμα. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω θα μπορούσε πράγματι να υπονομευθεί σοβαρά από τις τελευταίες εξελίξεις η σταθερότητα των τραπεζών η οποία είπατε ότι είναι καλύτερη που είχαμε ε, κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Ε, απάντηση. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που θέσατε, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητε, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, δηλαδή. Ε, πράγματι μας ανησυχούν ε, τα πολυάριθμα πρόσφατα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται ο τραπεζικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία βέβαια πλήττουν ακριβώ το κύρο του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματο. Ε, και βέβαια αυτό που θα πρέπει να ε, κάνουμε είναι να αντλήσουμε τα διδάγματά μα ε, και να αποκαταστήσουμε τις ζημιέ που έχουν προκληθεί. Ειδικότερα, εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πόσο ισχυρή είναι η ο εποπτικό μα έλεγχο. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό οι οδηγίε μα που έχουμε ακριβώ για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματο ε, εφαρμόζονται. Δηλαδή να δούμε στο πλαίσιο της εθνικής αρμοδιότητας, γιατί τα κράτη-μέλη είναι απόλυτα αρμόδια για την εφαρμογή ε, των λίγων οδηγιών, πώς γίνεται λοιπόν η εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ό,τι αφορά ακριβώς την ε, αξιολόγηση που προτείναμε των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στοχεύουμε ακριβώ αυτό. Δηλαδή να τους δώσουμε, να δώσουμε σε αυτές τις αρχές περισσότερες αρμοδιότητες έτσι ώστε να διασφαλίζουν την σωστή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρμοδίων αρχών έτσι ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν δράση σε περίπτωση που μία από αυτές τις αρχές διαπιστώσει ότι ε, υπήρξε μία παραβίαση αυτών των πρόσφατα συμπεφωνημένων κανόνων. Επίσης, ε, βρισκόμαστε τώρα σε μια ε, φάση συγκέντρωσης δεδομένων, ένα fact-finding δηλαδή, ε, προκειμένου ακριβώς να συγκεντρώσουμε στοιχεία για αυτά τα πρόσφατα, για τις ε, πρόσφατες περιπτώσεις κλιμάματος χρήματος, έτσι ώστε να διαφωτίσουμε καλύτερα αυτές τις περιπτώσεις και με βάση τα λόγω στοιχεία να δούμε ποιε είναι οι συμπληρωματικές δράσεις ε, που είναι απαραίτητες πέραν δηλαδή των, των τροποποιήσεων οι οποίες θα επέλθουν στο πλαίσιο της, του, της αξιολόγησης Μετά, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αντίκτυπο ενός ε, δυνητικού σκληρού Brexit στην ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη και ειδικότερα την σταθερότητα του συστήματος μας. Καταρχήν να πω πως ε, είναι ξεκάθαρο πως θα είναι ζημιογόνο από οικονομικής άποψης ένα σκληρό Brexit τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών. Γιατί βέβαια εδώ μιλάμε για δεκαετίε οικονομική ολοκλήρωση στην οποία συμπεριλαμβανόταν το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα. Εξετάσαμε ε, τα ζητήματα αυτά τα οποία είχε εντοπίσει η ομάδα εργασία που δημιουργήθηκε ανάμεσα στην Bank of England και την ECB. Ε, δηλαδή, ε, Τομεί εκείνου του οποίου θεωρούμε ότι υπάρξει ακριβώς κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα και ε, ακριβώς ε, εντοπίσαμε, αναγνωρίσαμε αυτού του τομεί και λάβαμε τα απαραίτητα μέτρα. Ωστόσο, σίγουρα δεν μπορούμε να αποτρέψουμε πλήρως ε, κάποιες απορριθμίσεις, κάποια προβλήματα που θα προκύψουν με ορισμένες επιχειρήσεις στην αγορά και γι' αυτό οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες έχουν ανακοινώσει και μέτρα διασφάλισης ρευστότητάς τους ε, και ακριβώς ε, την ε, θέση και πάλι σε, σε, σε λειτουργία αν θέλετε ενός ειδικού credit line ανάμεσα στην ECB και την Bank of England. Δεν νομίζω λοιπόν πως το ένα σκληρό Brexit πραγματικά θα μπορέσει να οδηγήσει σε σημαντική οικονομική μείωση, αλλά πραγματικά θα είναι σημειογόνο. Εκ μέρους των σοσιαλιστών τώρα, κ. Φερνάνδης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πριν από λίγα χρόνια το κόμμα μου δηλαδή, ε, με κάλεσε να συμμετάσχω ως υποψήφιο στις ευρωεκλογέ. Τότε ήταν δύσκολη απόφαση, γιατί έπρεπε να εγκαταλείψω την δικιά μου επαγγελματική ζωή στον ιδιωτικό τομέα. Ε, δέχτηκα ε, εξαιτία τη ιδεολογία. Επειδή κάποιο από εδώ μου είχε πει ότι η πολιτική σημαίνει να μαθαίνει κανεί να ζει με απογοητεύσει. Και η απογοήτευση είναι κάτι καθημερινό εδώ στο σώμα. Και τώρα που ολοκληρώνεται η θητεία μα, θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω για την απογοήτευση αυτή που ζούμε, επειδή καθυστερεί το έντις. Όπως ξέρετε, το Σώμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία. Και όχι γιατί έλειψε η βούληση από τη δικιά μου πολιτική ομάδα, και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω εσείς πώς βλέπετε τους επόμενους μήνες τα πράγματα, τι θα γίνει. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια συνάντηση για το χάρτη πορείας ε, στο Eurogroup. Εσείς τι πιστεύετε, υπάρχει περίπτωση να λυθεί μέρος τουλάχιστον του προβλήματος και να έχουμε λιγότερη απογοήτευση. Έπειτα με λιγότερη απογοήτευση έχουμε την ε, τιτλοποίηση των ΣΥΖΙΕΣ που όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί αλλά είμαστε εν αναμονή του Συμβουλίου και νομίζετε το Συμβούλιο έχει όρεξη να το προχωρήσει. Γι' αυτό τα δύο θέλω λοιπόν να σας ε, ρωτήσω έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η θητεία με κάπως λιγότερη απογοήτευση από αυτήν που έχουμε συγκεντρώσει σήμερα. Απάντηση. Τι μπορώ να πω για αυτά. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο και εγώ την ίδια απογοήτευση νιώθω. Αν κοιτάξετε τι έχει γίνει με το έντις, η πρόοδος είναι ελάχιστη. Και ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει χάρη στην δική σας επιτροπή, την κυρία Λάγκε, την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Τον Νοέμβριο του 2016 ξεκίνησε η υπόθεση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πετύχει πολιτική πρόοδο και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ δεν θα υπάρξει καμία πρόοδος πριν από τις επόμενες ευρωεκλογέ. Γίνεται βέβαια δουλειά σε τεχνικό επίπεδο, αλλά δεν μπορέσαμε πολιτικά να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Συνεπώς, το μόνο θετικό νέο είναι ότι το έργο αυτό δεν έχει σταματήσει πλήρως. Υπάρχει ομάδα υψηλού επίπεδου για το ΕΝΤΙΣ που εργάζεται στο Συμβούλιο. Βέβαια, δεν λέω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την διακυβερνητική προσέγγιση. Και τι να πω, ίσως αν είχε υπάρξει περισσότερη σύγκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είχαν ξεκινήσει πολιτικές συζητήσεις και στο Συμβούλιο. Πάντως, από τότε που έγινε η πρόταση αυτή τον Νοέμβριο του 2015 έγιναν και πάρα πολλές προσπάθειες για την μείωση κινδύνου και αναφερθήκαμε σε αυτές. Ορίμασε πια η κατάσταση για να προχωρήσουμε και στον επιμερισμό κινδύνου και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το έργο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως να υπάρχει κάποια δυνατότητα με το ΕΣΠΙΣ. Γιατί το Συμβούλιο δεν προχώρησε μέχρι τώρα και με την Αυστριακή Προεδρία που αποφάσισε να μην προχωρήσει περισσότερο με την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Αυστριακή Προεδρία. Αλλά αυτό που είναι θετικό τώρα είναι ότι έχει συμφωνηθεί η έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής. Θα ψηφίσετε από ό,τι κατάλαβα 15 Απριλίου στο Στρασβούργο. Άρα θα φανεί ότι υπάρχει ο φάκελος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να προχωρήσει και μια που υπάρχουν συζητήσεις και όσον αφορά το έντις για τα ανοίγματα κρατικών ομολόγων αυτό είναι μια δυνατότητα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο στο θέμα αυτό των κρατικών ομολόγων και το άνοιγμά τους. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να δουλεύουμε και ελπίζω να ε, τα καταφέρουμε. Σημερίζουμε την απογοήτευσή σας. Δεν πρέπει να παραιτηθούμε όμως και ελπίζω στην επόμενη θητεία να συνεχιστεί το έργο μας. Ευχαριστούμε. Πάλι ΕΛΚ. Μάρκος Φέμπερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν νομίζω πως θα εκλαγείτε πολύ αν για το ΜΥΦΙ 2, αλλά γνωρίζουμε ως, ότι ως το Μάρτιο του 2020 η Επιτροπή θα πρέπει να προετοιμάσει μία έκθεση σε ό,τι αφορά τις διάφορες επιτυχίες των υποχρεώσεων που προβλέπει το MIFID 2. Αλλά η ΕΣΜΑ έχει προβεί σε μία δήλωση, την οποία βρήκα στην ιστοσελίδα της, ότι ε, το input, δηλαδή τα στοιχεία ε, για αυτή την έκθεση που θα πρέπει να συντάξει η Επιτροπή, ε, θα διατεθούν από την πλευρά της ε, ΕΣΜΑ με καθυστέρηση 6 έως 24 μηνών. Αυτό τουλάχιστον διάβασα από την πλευρά της, ΕΣΠΑ, οπότε θα ήθελα, ε, ΕΣΜΑ, οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, ήρθατε σε επαφή με την ΕΣΜΑ. Μπορεί να δώσει κάποιες διευκρινήσεις, μπορεί να ανταποκριθεί στι προθεσμίε που είχαμε προβλέψει. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει εργασίε οι δικέ σα εσωτερικά στην Επιτροπή, γιατί βέβαια πλησιάζει το 2020, δεν απέχει πολύ ακόμα. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά. Τις ερωτήσεις σας για το Μηφίδιο. Ναι, πράγματι στις 27 Μαρτίου η ΕΣΜΑ ε, δημοσίευσε μια επιστολή, επιστολή που ευθύνεται στην Επιτροπή, στην οποία προτείνει μία αναβολή κατά 6-24 ε, μήνες των ε, αξιολογήσεων σε ό,τι αφορά το MIFID 2020 που για το που έχουν προβλεφθεί ακριβώς λόγω του, του ενδεχόμενου Brexit η δική μας αντίδραση είναι ότι δυστυχώς η ΕΣΜΑ δεν θα προβεί ακριβώς στην διάθεση των σχετικών στοιχείων εγκαίρως. Αλλά από την άλλη πλευρά ισχύει το ότι για να γίνει η ανάλυση και να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις θα πρέπει να υπάρξει και ακριβώς μια σαφήνεια ως προς το πώς θα διαμορφωθεί το, η εμπορική αν θέλετε, κατάσταση, γενικότερα η κατάσταση οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη σε περίπτωση ενός Brexit. Και ε, ε, η σχετική πρόταση όταν ό,τι αφορά την ενοποιημένη έκθεση η οποία θα, αποσ... Ε, η οποία θα προετοιμαστεί ήδη και το σχετικό αίτημα δηλαδή προς την ΕΣΜΑ είχαν σταλεί από τη δική μας ε, πλευρά εγκαίρως προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την ε, έκθεση του 2020. Ε, είδα βέβαια πως, ο πρώτος, έχει προσέρθει ο κ. Λάγκη, αλλά κυρία Βέντερ έχετε το λόγο εσείς τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα λοιπόν και εγώ από την δική μας πλευρά. Είσαστε αρμόδιος αντιπρόεδρο και επίτροπο δηλαδή, ε, για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο. Οπότε θα ήθελα να σα θέσω ένα ερώτημα προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, στο πλαίσιο λοιπόν των διάφορων ε, ε, πακέτων διάσωση και της, των πολιτικών λιτότητα που είδαμε κατά την τελευταία περίοδο, τα ζητήματα εθνική κυριαρχία βέβαια τέθηκαν καθώ υπήρξαν και τριβέ σε ό,τι αφορά τον τομέα τη κοινωνική διασφάλιση. Και μέσα σε όλο αυτό βέβαια έχασε κατά κάποιο τρόπο σε κύριο, σε φήμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε, στο πλαίσιο αυτή τη ε, ολοκλήρωση τη βουλευτική ε, ε, θητείας, ποια θεωρείτε πως ήταν τα επιτέματα, ποια ήταν τα ορόσημα τα οποία καταφέραμε στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και τι κάναμε δηλαδή ω προσπάθειες ούτω ώστε ακριβώ να υπάρξει ένα καλύτερο συμβιβασμό μεταξύ του κοινωνικού διαλόγου Αφενό και ε, του ευρώ γενικότερα αφετέρου. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, ένα ζήτημα που έθεσε και λίγο προηγουμένω ο συνάδελφο Σιβέν Γκίγκολτ, να πω ότι ακριβώ αυτή η βιωσιμότητα σχετίζεται και με την κοινωνική διάσταση, δηλαδή ε, την διασφάλιση κοινωνικών προϋποθέσεων αλλά δυστυχώ σε ό,τι αφορά τι προτάσει που κάναμε εμεί ω σοσιαλιστέ, σε ορισμένε περιπτώσει αποτύχαμε. Δηλαδή δεν συγκεντρώσαμε τι αντίστοιχε πλειοψηφίε. Οπότε θα θέλαμε να σα ρωτήσουμε, θεωρείτε πω υπάρχει ακριβώ ανάγκη να λαμβάνετε και η κοινωνική διάσταση περισσότερο υπόψη σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα των επενδύσεων και πώ θέλετε να το αντιμετωπίσετε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα. Σε ό,τι αφορά το πιο γενικό ερώτημα που θέσατε, σε ό,τι αφορά ε, την κοινωνική διάσταση και το τι έχουμε κάνει στο πλαίσιο της ε, τρέχουσας ε, επιτροπής και το ποια είναι τα, τα ορόσημα εκείνα, τα επιτεύγματα τα οποία θα μπορούσα να αναφέρω, να σας πω ότι πράγματι η δική μας επιτροπή έχει κάνει προσπάθειες ώστε να προωθήσει την κοινωνική ατζέντα κοινωνικό θεματολόγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα ορόσημο που θα μπορούσα να αναφέρω είναι ο Ευρωπαϊκός Επιλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ο οποίος συμφωνήθηκε και σε συνέχεια του οποίου ήρθα μία σειρά από νομοθετικές προτάσεις από την πλευρά της Επιτροπής, για παράδειγμα, ε, κοινωνική προστασία για όλους και προσαρμογή των κανονισμών που έχουμε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον, ε, την αγορά εργασία, ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στι ε, διαφορετικέ μορφέ εργασία που έχουν ε, ανακύψει. Και εδώ πάντοτε έχουμε ως στόχο ε, του, να, του ανεξαρτήτως του ποιο είναι, ποια είναι η σύμβαση εργασίας, είτε μιλάμε για αυτό απασχολούμενο, μερικώς απασχολούμενο, πλήρως απασχολούμενο, να υπάρχει η κατάλληλη κοινωνική προστασία της οποίας θα χαίρει ο εργαζόμενος. Αυτό λοιπόν μπορώ να σας αναφέρω σε ε, παράδειγμα, ε, δηλαδή ε, τη συνέχεια που δώσαμε στον κοινωνικό πυλώνα και από εκεί και μετά έχουμε και το ευρωπαϊκό εξάμεινο και το 30% των σχετικών κοντιλίων τα οποία σχετίζονται του ευρωπαϊκού εξάμεινου με ακριβώς με ζητήματα της αγοράς εργασίας. Και κατά τελευταία δύο χρόνια όταν ε, ε, συζητούσαμε τις προτεραιότητες της οικονομικής ε, πολιτικής σε ό,τι αφορά επενδύσεις, σε ό,τι αφορά διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, πάντοτε δίναμε έμφαση στην διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης για όλους και της μείωσης των ανισοτήτων εδώ, σε ό,τι αφορά το εισόδημα. Τώρα, έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα που θέσατε, σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα των επενδύσεων. Καταρχήν να σας πω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να υιοθετήσει μια σφαιρική, μια ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα και προκειμένου δηλαδή να ε, λαμβάνει υπόψη και ε, όλους τους ε, παράγοντες, δηλαδή κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και ό,τι καθεξής. Σε ό,τι αφορά Σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση, προφανώ δώσαμε έμφαση και στην περιβαλλοντική διάσταση, γιατί είπαμε ότι υπάρχει εδώ προτεραιότητα, υπάρχει επίγοντο χαρακτήρα και θα πρέπει να ανταποκριθούμε και στι ε, υποχρεώσει και τι δεσμεύσει που αναλάβαμε στο πλαίσιο Συμφωνία των ε, Παρισίων. Αλλά στην ίδια ε, πρόταση περιλαμβάνονται και ελάχιστα κοινωνικά, ε, κοινωνικές δικλείδες ασφαλείας, αν θέλετε. Και είμαστε διατεθειμένοι να ε, διευρύνουμε αυτές τις εργασίες ε, και να δημιουργήσουμε και περαιτέρω ταξινομήσεις. Δηλαδή ξεκινώντας από το περιβάλλον αλλά στη συνέχεια πηγαίνοντας και στον τομέα της διακυβέρνησης και στον τομέα ακριβώς των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Και χαιρετίζουμε την, την αναλογική, αν θέλετε, ευρωσέγγιση που ακολουθεί και η κοινή επιτροπή σε ό,τι αφορά τις ταξινομήσεις αυτές. δεν έχει ακόμα ασχοληθεί με την ε, ταξινόμηση σε ό,τι αφορά τα, ε, τις κοινωνικές επιτυχίες, αλλά στο πλαίσιο ακριβώς της συνέχισης των εργασιών έχει αναλυφθεί αυτή η δέσμευση, ότι δηλαδή θα εξεταστεί και η κοινωνική ταξινόμηση. Και ο Στέφαν Γκέρολτος, τελευταίος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για την παρουσίαση που μας κάνατε. Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά αυτήν την ε, ταξινόμηση σε ό,τι αφορά την, ε, τα, τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, το sustainable financing. Ε, εκείνο που εγώ δεν μπορώ να, να, να, διασφαλίσω, αν θέλετε, με αυτή την ταξινόμηση ότι μπορεί να αποφέρει υψηλά έσοδα, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο ε, προϊόν. Γιατί πώς μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο ε, κάτι τέτοιο για ένα προϊόν το οποίο δημιουργεί ένα είδο ε, κινδύνου για τον επενδυτή σε αυτό. Πώς μπορεί λοιπόν ε, η Επιτροπή να διασφαλίσει σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν ζήτησε και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι ένας επενδυτής δεν θα προβεί στην επένδυση σε ένα λανθασμένο προϊόν. Περίπλοκη αυτή η ερώτηση, λέει ο κ. Και χρειάζεται ευρύτερη απάντηση. Βεβαίως η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά ε, εργαλεία ή προϊόντα ε, ενέχει κινδύνους ε, διαφορετικά εργαλεία ή προϊόντα μπορεί να ενέχουν διαφορετικούς κινδύνους και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και μάλιστα κατά την έννοια αυτή έχουμε αναλάβει και κάποιες ε, πρωτοβουλίες έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι επενδυτές, οι καταναλωτές ε, είναι προετοιμασμένοι κυρίως ε, οι επενδυτές καταναλωτές λιανικής να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι για τους κινδύνους που σχετίζονται με οποιαδήποτε χρηματοδοτικά, χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Ε, όσον αφορά τα πράσινα επενδυτικά προϊόντα. Ε, κανένας δεν λέει ότι αυτά δεν θα έχουν κανένα βαθμό κινδύνου. Είναι επίσης ε, χρηματοπιστωτικά εργαλεία, προϊόντα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι και μέσω αυτής ε, της ε, ταξονομίας ότι υπάρχει η απαραίτητη σήμανση, η θέσπιση ε, προϋποθέσεων και κριτηρίων κτλ. και ε, ε, λέμε ότι πρέπει τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα όσον αφορά αυτά τα βιώσιμα προϊόντα και πρέπει να υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ε, αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα ε, παρουσιάζονται. Αυτά όσον αφορά το βιώσιμο σχέδιο ε, δράσης. Εκεί τα συζητήσαμε και τα benchmarks και όλα. Και την, αυτή την ταξινόμηση. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που αφορούν και εμπίπτουν μάλλον στους γενικότερους ρυθμιστικούς μας ε, κανόνες. Το Catch the Eye τώρα. Ο κύριος Λάγκεν πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Στην αρχική παρουσίαση που κάνατε αναφέρεται μια σειρά από εξετάσει ε, που κάνατε και μεταρρυθμίσει που ξεκινήσατε και πραγματικά πρέπει να πω ότι έγινε δουλειά από πλευρά τη Επιτροπή. Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε. Πάντω, στην αρχή τη ε, θέτια αυτής είχε ε, προβλεφθεί μια συνολική, μια σφαιρική αξιολόγηση όλου του κανονιστικού πλαισίου για τι τράπεζε, λαμβάνοντα υπόψη και το διεθνέ πλαίσιο, δηλαδή συγκρίνοντας τη, τη διεθνή κατάσταση και κάνοντα μια αντιπαραβολή μεταξύ μικρών τραπεζών και μεγάλων τραπεζών. Δηλαδή, στην Αμερική η αντίστοιχη ορολογία είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο για το Main Street και ένα κανονιστικό πλαίσιο για το Wall Street. Οπότε θα ήθελα να σας πω εσείς σε ποιο βαθμό έχετε ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση. θα προλάβετε, επειδή είχατε αναφέρει ε, τον Οκτώβριο ότι θα προβείτε σε μια τέτοια συνολική αξιολόγηση του τι έχουμε επιτύχει, ε, θα προλάβετε να το κάνετε στο πλαίσιο της δικής σας θητείας ακόμα κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κατά μια έννοια, είχαμε ήδη μια τέτοια σχέση. Είναι η αίτηση για στοιχεία και δεχτήκαμε ότι βεβαίως η προηγούμενη εκθέση είχε προετοιμαστεί ε, βιαστικά λόγω της ε, κρίσης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τώρα βλέπουμε ε, που έχουν υπάρξει επικαλύψεις, που έχουν προκύψει ελλείψεις. που υπάρχουν κενά ή κάποιες ε, μη επιθυμητές ε, επιπτώσεις κλπ. Δουλεύουμε επί της βάσεως αυτής. Και δίνουμε σάκα και οστά κατά κάποιο τρόπο ε, σε αυτές τις ε, μαρτυρίες ε, μέσα από νομοθετικά κείμενα, το ρέφιτ κλπ. Να σας πω ότι μία από τις δράσεις follow-up είναι ένας έλεγχος κατάστασης fitness check όσον αφορά ε, τη διαδικασία ε, reporting. Έχει δουλέψει η Κομισιόν πάνω σε αυτό το θέμα έτσι ώστε να δει την αποτελεσματικότητα ε, της εποπτείας όσον αφορά την κατάσταση της αγοράς και την εποπτεία των διαφόρων προϊόντων έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα προαπαιτούμενα ε, είναι σωστά ε, και βεβαίως αυτή η έλεγχη ε, fitness check, έλεγχη κατάστασης πρέπει να έχουν και μία μακρόθωρη ας πούμε δράση και βεβαίως μετά θα δούμε ε, και ποιες ε, είναι οι δυνατότητες απλούστευσης ε, του, της διαδικασίας αναφοράς του reporting, αλλά αυτά θα πρέπει να τα κάνει η επόμενη Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αναφερθήκατε, απαντώντας στον συνάδελφο Φερνάντες, τον φάκελο Έντις. Να σας πω ότι ο προκάτοχός σας Μάλλον η κυρία Κιόνιγκ που καθόταν στη θέση σας πριν ε, μας είπε ότι το καλύτερο μοντέλο ήταν το Αμερικάνο του FDIC και όχι η ανακοίνωση που μας ε, κάνατε στην ενδιάμεση εξέταση του θέματος. Ίσως ε, θα πρέπει να πείτε, ε, να προτείνετε στους επόμενους από εσά μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση. Όσον αφορά το MIFID, μετά από το Brexit, τι γίνεται. Τώρα, αν η ΕΣΜΑ θέλει να δουλέψει τώρα ή αργότερα είναι ένα θέμα. Το άλλο ζήτημα είναι πώς φαντάζεστε εσείς να γίνεται αυτή η αναθεώρηση. Αυτή τη στιγμή ε, ε ξέρουμε ότι υλοποιήθηκε όλη αυτή η διαδικασία όταν ε, ε, βρίσκονταν πλήρως στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η, η Βρετανική Κεφαλή Αγορά θέλετε να μας πείτε ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές ε, της ε, επίπτωσης του Brexit στο MIFID, γιατί νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί απλά μια μικρή τεχνική αναθεώρηση όπως είχε υποθεί αρχικά. Ποιες θα είναι οι κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές ε, τις οποίες θέλετε να ακολουθήσετε πέρα και έξω από, τις, από τα τεχνικά δελτία. όσον αφορά το έντις ε, και για να επανέλθουμε στο ίδιο ζήτημα. Ναι, μπορεί η Έλκα να έκανε διαφορετικά σχόλια. Εγώ δεν μπορώ να ευθυγραμμιστώ απαραίτητα ε, για το έντις. Επί της ουσίας δεν μπορεί να αλλάξει η θέση μας. Είναι ένα ε, σφάκελος επί του οποίου η πρόοδος ή το αργεί. Από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι οι πυλώνες, της επιτήρησης, ε, οι είναι επιτήρηση, εξυγίανση ε, και διασφάλιση καταθέσεων και επομένως εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την προσέγγιση μέσω των τριών πυλώνων βεβαίως εάν στην διαβούλευση με τα κράτη-μέλη και με τη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκύψει κάτι άλλο, μια διαφορετική προσέγγιση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική συμφωνία, τότε ναι φυσικά θα είμαστε απολύτως διατεθειμένοι να διερευνήσουμε αυτές τις νέες προτάσεις. Ε, κατά μία έννοια έχουμε ήδη κάνει κάτι παρόμοιο το το φθινόπωρο του 17, αν δεν κάνω λάθος, είχε υπάρξει μια ανακοίνωση παρατήρηση εκτό μικροφώνου τη κυρίας Μπερές. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος, αυτό μπορεί κανείς να το συζητήσει. Εν πάση περιπτώσει αποτέλεσε μια προσπάθεια απεμπλοκή ε, τη ε, συζήτηση. Ναι, δεν ε, είχε αίσιο τέλος αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που τουλάχιστον δεν έχει μπλοκάρει τελείως η κατάσταση. Ε, αποτέλεσε μια προσπάθεια διευκόλυνση του πολιτικού συμβιβασμού. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε αν και κατά πόσον μπορούμε να διερευνήσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην πολιτική συμφωνία. Όσον αφορά τώρα το θέμα του MIFID και την αναθεώρηση του MIFID, πού τα έχω τα χαρτιά μου τώρα. Να τα ψάξω. Α, τα βρήκα. Αναθεώρηση MIFID. Επί του παρόντος ε, βρισκόμαστε σε φάση προετοιμασίας. Πριν από 18 μήνες άρχισε να λειτουργεί ε, η οδηγία, επομένως μπορούμε να εξάγουμε κάποια διδάγματα ήδη. Το θέμα προστασίας των καταναλωτών είναι πολύ σημαντικό ε, καθώς επίσης ε, και η λειτουργία των μετοχών και των ε, ομολόγων. Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα για μεγαλύτερη διαφάνεια αγοράς και όπως είπα και προηγουμένως θέλουμε αυτές οι εκθέσεις να απασχολήσουν κατά προτεραιότητα την ΕΣΜΑ. Επίσης, αυτή τη στιγμή ε, ε, κατά πόσον έχει λειτουργήσει ε, καλά ο διαχωρισμός του broking από, τις, από την αξιολόγηση επενδύσεων κυρίως ε, για ε, όσον αφορά τις μικρές μεσαίες ε, επιχειρήσεις. Αυτές είναι κάποιες από τις κατευθύνσεις της εργασίας μας όσον αφορά αυτήν την αναθεώρηση. Και τώρα τελευταία ερώτηση από τον κύριο Τρεμόσα. Ευχαριστώ πολύ. Για τις τέσσερις μεγάλες. Σήμερα στα Financial Times υπάρχει ένα άρθρο που λέει ξυπνήστε τους τέσσερις μεγάλους και φροντίστε να τους υποβάλλετε στη... στους προληπτικούς ελέγχους. Εσείς πρόσφατα απαντήσατε σε γραπτή δική μου ερώτηση πριν από μερικούς μήνες και είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την αγορά ελέγχου ώστε να τηρείται η νομοθεσία που έχει ήδη υιοθετηθεί από το 2014. Αλλά λέτε ότι υπάρχουν χώρες που ακόμα δεν έχουν ενσωματώσει τη νομοθεσία την ευρωπαϊκή. Μπορείτε να ξέρουμε λοιπόν ποιες είναι οι χώρες αυτές οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει την νομοθεσία που εγκρίθηκε πριν από πέντε χρόνια και δεν την έχουν ενσωματώσει ακόμα στην εθνική τους νομοθεσία. Μάλιστα, απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όσον αφορά τους τέσσερις μεγάλους, έχουμε την λογιστική μας ρύθμιση. Δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η ακριβής κατάσταση ενσωμάτωσης. Δεν έχω την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την ενσωμάτωση της οδηγίας αυτής στην εθνική νομοθεσία. Θα μπορούσα ίσως να ζητήσω από τους συναδέλφους να σας απαντήσουν. Πάντως παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην αγορά. Και αυτό σύμφωνα με τα ρυθμιστικά πλαίσια που διαθέτουμε. Αυτό μπορώ να σας πω τώρα. Πάντως θα παρακολουθήσουμε και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό της ενσωμάτωσης της οδηγίας στην Εθνική Νομοθεσία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Όντως ήρθατε εδώ υπό μία από τις ιδιότητές σας, ίσως σας ξαναδούμε σύντομα. Και ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους για την συμμετοχή τους. Διακόπτουμε για πέντε λεπτά και μετά θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και εκτιμούμε όλο ιδιαίτερος τη μια μισή ώρα που καθίσατε εδώ μαζί μας κύριε Αντιπρόεδρε. Oh, oh. Okay. Okay. Okay, so we just continue, sir. Okay. Thanks. Good luck. So they said want to continue. So this was the problem. That was the point. Yeah, okay.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

Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σας διάταξης, σημείο 21. Οπότε, εξετάζουμε τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και περνάω στα αγγλικά, λέει η κυρία Μπερές, που είναι στη θέση της Προέδρου. Πρόκειται για μελέτη της ΕΚΟΝ όσον αφορά τα εφαρμοστικά μέτρα και τις κατεξοδότηση πράξης. Είναι τελευταία φορά σε αυτή τη θητεία και εμείς κάθε φορά λέμε ότι η Οικονομική Επιτροπή δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις ε, εποπτικές της αρμοδιότητες, μερικές φορές για πολύ περίπλοκες πράξεις. Πιστεύουμε ότι η δημόσια συζήτηση είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να εκτιμήσει την ε, προληπτική αρμοδιότητα σωστά και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Η σημερινή συζήτηση επικεντρώνεται στην αναθεώρηση των ε, εκτελεστικών μέτρων όσον αφορά την Οδηγία 2009-188 προκειμένου να συνεχίσουμε το έργο μας όσον αφορά τις ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις. Υπάρχει και τροπολογία για κατεξοδότηση πράξη όσον αφορά την αναθεώρηση διαφόρων στοιχείων της ε, Φερεγγιότητα 2 και τις κεφαλαϊκές απαιτήσει μετά από ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τροπολογίες και το έργο της ΑΙΟΠΑ στο τομέα της δημόσιας διαβούλευσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά υιοθέτησε την τροποποιημένη πράξη Solvency 2 στις 28 Μαρτίου προκειμένου να συζητηθούν οι τροπολογίες αυτές σήμερα καλωσορίζω εδώ τον κύριο Μερλά εκ μέρου της Digifisma και τον κύριο Ρέι εκ μέρου της ΕΙΟΠΑ της Ευρωπαϊκή Αρχής Ασφάλιση και Επαγγελματικών Συντάξεων. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μερλά πρώτα απ' όλα για να μας παρουσιάσει την αναθεώρηση αυτή της καταξιδότηση πράξης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη αυτή τη Επιτροπή. Ε, Σα καλημερίζω. Όπω γνωρίζετε, η οδηγία Περιγκιότητα 2 άρχισε να ισχύει στι αρχέ του 2016 και η συμφωνία ε, για αυτή την οδηγία και για την εφαρμογή της ε, χρειάστηκε την, μεγάλες προσπάθειες από την πλευρά του κλάδου, των αρμόδιων για τη χάραξη της πολιτικής και των νομοθετών και θεωρούμε πως οι προσπάθειες αυτές τελικά απέφεραν καρπούς καθώς ε, η θέσπιση αυτού του νέου πλαισίου για την προληπτική εποπτεία πήγε αρκετά καλά. Ε, παρότι δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο, παρόλα αυτά η οδηγία, αυτή η Φερεγγιότητα 2, ε, εισήγαγε μια σειρά από καινοτόμα στοιχεία και έχει προβλεφθεί και μια σειρά από εξολογήσει ε, ε, ε, το 2020 θα προβούμε σε μια ευρεία επαναξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας ενώ αυτή την περίοδο εξετάζουμε ε, και αξιολογούμε τα εφαρμοστικά μέτρα. Αυτή λοιπόν η αξιολόγηση μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα σχόλια που λάβαμε στο πλαίσιο του Call for Evidence, δηλαδή της πρόσκλησης για την υποβολή στοιχείων που κάναμε το 2015 και επίσης θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε περαιτέρω πρόοδο σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας ένωσης κεφαλαίου αγορών. Και προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν η Επιτροπή αναγνώρισε τρεις ε, τομεί στους οποίους εστίασε. Πρώτον, η αναλογικότητα. Δεύτερον, η αφαίρεση, η εξάλληψη, αν θέλετε, αθέλητων τεχνικών ασυνεπιών και τρίτον, η αφαίρεση των εμποδίων για τις επενδύσεις. ο αναθεωρημένος τώρα κατεξοδότηση κανονισμός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 8 Μαρτίου και περιλαμβάνει βελτιώσεις και καλύτερη ευθυγράμμιση ανάμεσα στην ε, νομοθεσία του ασφαλιστικού και του τραπεζικού τομέα, περισσότερη αναλογικότητα σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αποτήσεων, διατάξει σε ό,τι αφορά τη λήψη υπόψη των πρόσφατων εξελίξεων στην διαχείριση του κινδύνου, αλλαγές σε ό,τι αφορά την διαδικασία του, ε, του καθορισμού ε, των επιτοκίων ε, χωρίς κίνδυνο της ώστε να αντιπακρονόμαστε καλύτερα στις νομικές αρχές και επίσης περιλαμβάνει και ενημερώσεις σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις, σε ό,τι αφορά ορισμένα ανοίγματα προκειμένου να απηχεί καλύτερα πιο πρόσφατα δεδομένα. Αυτές λοιπόν οι στοχευμένες τεχνικές αλλαγές θα διασφαλίσουν ότι η οδηγία Φεραγκαιότητα 2 παραμένει επίκαιρη. Στον τομέα των επενδύσεων έχουμε βελτιώσει την μεταχείριση των ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων και των ιδιωτικών τοποθετήσεων χρέου, ε, ανταποκρινόμενα σε κριτήρια τα οποία είχαν ε, προταθεί από την ΕΙΟΠΑ στην ε, γνωμοδότησή της. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις αλλαγές ε, θα ε, συμβάλλουμε στην δημιουργία πιο δραφοροποιημένων πηγών χρήματοδότηση για την πραγματική οικονομία. Μετά από το τελευταίο λοιπόν scrutiny slot, δηλαδή την τελευταία εξέταση ε, και μετά από την επιστολή που στείλατε στον ε, Αντιπρόεδρο τον Πρόφστη στο Σεπτέμβριο αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε και μια πιο εξατομικευμένη μεταχείριση των μακροπρόθεσμων μετοχικών κεφαλαίων παρότι δεν είχαμε ζητήσει σχετική συμβουλή από την ΕΙΟΠΑ. και με αυτή την νέα τώρα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων θα ε, τις εξασφαλίσουμε και μια χαμηλότερη κεφαλαιακή επιβάρυνση στις τάξη του 22%. Ό,τι δηλαδή ισχύει και για τις στρατηγικού χαρακτήρα συμμετοχές. Ε, το σχετικό σχέδιο για την κατεξοδότηση πράξη δημοσιεύθηκε στο πόρταλ για την καλύτερη νομοθεσία στις 9 ε, Νοεμβρίου και λάβαμε 25 απαντήσεις από τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Ε, και εξετάσαμε τα εν λόγω σχόλια κατά τις τελευταίες εβδομάδες και κάναμε μία σειρά από προσαρμογές στην, στο αρχικό μας κείμενο. Καταρχήν, μία σειρά από φορεί ε, σχολίασαν τα κριτήρια για τη νέα κατηγορία των μακροπρόθεσμων, δηλαδή μετοχικών κεφαλαίων, ε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την, ελάχιστη, την απέτηση τη ελάχιστη περίοδου παρακράτηση των 12 ετών ε, και το κριτήριο του ring fencing, τη κλειστή διάρθρωση. Προκειμένου λοιπόν να λάβουμε υπόψη μα αυτά τα σχόλια, αποφασίσαμε να μειώσουμε πολύ σημαντικά την προπόθεση ακριβώ την απέτηση σε ό,τι αφορά την ελάχιστη παρακράτηση. Τη μειώσαμε σε 5 χρόνια και αφαιρέσαμε επίση οποιαδήποτε αναφορά στο ring fencing, στην κλειστή διάρθρωση. Επίσης θα ε, αναβάλουμε την ημερομηνία εφαρμογής ε, των νέων απαιτήσεων σε ό,τι αφορά ε, την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλόμενων φόρων για αρχέ στις αρχές του 2020. Έτσι λοιπόν ο κλάδος θα έχει περισσότερο, χρόνο για να εφαρμόσει τους νέους κανόνες της ε, προληπτικής εποπτείας. Επίσης αποφασίσαμε να διευκολύνουμε την εφαρμογή της ε, προτιμησιακής μεταχείρισης ό,τι αφορά μη διαβαθμισμένους χρωστικούς ε, τίτλους, όπου δηλαδή οι ασφαλιστές επενδύουν μαζί με τράπεζες και άλλους ασφαλιστές. Και έχουμε μειώσει το απαιτούμενο ποσοστό παρακράτησης για τον συνεπενδυτή, για τον δεύτερο επενδυτή, από 50% σε 20%. Γνωρίζουμε με τις θέσει τώρα που έχει εκφράσει η δική σα Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εργοποίηση του εθνικού τμήματος της προσαρμογής μεταβλητότητας και του περιθωρίου ε, κινδύνου. Σε ό,τι αφορά τώρα την προσαρμογή ε, της μεταβλητότητας ε, χαιρετίζουμε ε, την βραχυπρόθεσμη λύση που βρέθηκε από τους συνομοθέτες στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, του FCF. Και η προσπάθεια ό,τι αφορά την εξέβραση μιας μακροπρόθεσμης σωστής λύσης θα συνεχίσουν στο πλαίσιο τη προετοιμασία τη αξιολόγηση του 2020. Σε ό,τι αφορά τώρα το περιθώριο κινδύνου, έχουμε λάβει εκτενεί συμβουλέ από την ΕΟΠΑ ότι ε, δεν είναι δικαιολογημένη μία μείωση του, ε, της κεφαλαιακής επιβάρησης ε, και κατά συνέπεια η επαναξιολόγηση που θα γίνει της οδηγίας δηλαδή της Φεραγιότητας 2 το 2020 θα μας επιτρέψει να επαναξετάσουμε γενικότερα αυτό το ζήτημα. Αυτή η αξιολόγηση του 2020 επίσης θα επιτρέψει την εις εξέταση γενικότερα τη οδηγία Φερεντιότητα 2. Και σε αυτό το πλαίσιο ήδη αποστήλαμε μια ε, ευρεία πρόσκληση για την υποβολή σχολείων στην ΕΙΟΠΑ που καλύπτει 19 διαφορετικού τομέου. Και επίση ζητούμε από την ΕΙΟΠΑ να προβεί σε μια ε, σφαιρική, μια πλήρη επαναξιολόγηση των ε, διαφόρων μέτρων εξασφάλιση των guarantee measures συμπεριλαμβανομένη τη προσαρμογή μεταβλητότητα και επίση ζητούμε την ΑΙΟΠΑ να κάνει προτάσει έτσι ώστε να ε, απηχούν καλύτερα τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των δραστηριοτήτων στον ασφαλιστικό τομέα σε ό,τι αφορά τι κεφαλαιατικέ απαιτήσει. Ήδη το Σεπτέμβριο του 2018 ζητήσαμε από την ΕΟΠΑ να ε, προβεί σε μια γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά ε, τον αντίκτυπο των κανόνων της, του εποπτικού ελέγχου για τι ασφαλιστικέ επιχειρήσει σε ό,τι αφορά τι βιώσιμε επενδύσει με βάση και το σχετικό σχέδιο δράσης τη Επιτροπής. Και επίσης εμείς θα ενημερώσουμε βέβαια ε, την ε, σχετική ε, έκθεση της Επιτροπής με βάση αυτά τα στοιχεία που θα λάβουμε και την οποία έκθεση τη δική μας θα την παρουσιάσουμε στους συνομοθέτες το 2020. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της ΕΙΟΠΑ. Έχετε 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής μετά από αίτημα της Επιτροπής για παροχή τεχνικών συμβούλων όσον αφορά ε, τον ε, κανονισμό ε, για την Αφαιρεγγιότητα 2, πρέπει να σας πω ότι η ΕΟΠΑ αντιμετωπίζει το θέμα βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και ε, με το μέλημα της εξασφάλισης της ε, ανα, ε, αναλογικότητας καθώς επίσης και κάποιες άλλες επιστοποιήσεις που οδηγούν στην τεχνική ε, ολοκλήρωση καθώς επίσης ε, και την επαναστοχοθέτηση οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ε, διαφορετική και διαφορετική κεφαλιακή επιβάρυνση όσον αφορά την όσον αφορά την, την οικονομική σταθερότητα. Ε, εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερως ε, τις ε, τροπολογίες τις οποίες η Επιτροπή σας έχει λάβει υπόψη της και είναι πολύ θετικές σε σχέση και με την θέση της ΕΙΟΠΑ. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υπάρχουν προβλήματα όπως είναι η, προσαρμογή της μεταβλητότητας, ε, καθώς επίσης και οι διαφορετικές, ε, τα διαφορετικά επιτόκια κλπ. Ε, ο, επίσης η ΕΟΠΑ συστήνει την τροποποίηση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά το sub-module του κινδύνου που παρουσιάζουν τα ποσοστά, τα επιτόκια. Αυτό η, η πρότασή μας είναι να ε, διορθωθούν ε, οι ελλείψεις ε, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να υλοποιηθούν. Λυπούμεθα γιατί η πρόταση αυτή, η δικιά μας πρόταση δεν φαίνεται καθαρά στις τροπολογίες του κανονισμού. Παρόλα αυτά σε γενικές γραμμές μπορεί να είναι σωστή η τοποθέτηση. Όσον αφορά το equity risk, οι τροπολογίες στον κανονισμό συμπεριλαμβάνουν και τη μείωση της κεφαλιακής επιβάρυνσης όσον αφορά αυτές τις επενδύσεις με μία περίοδο διακράτησης 5 ετών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, η αφαιρεγγιότητα 2 αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο ε, ε, της επαναδιαπραγμάτευσης της κεφαλιακής επιβάρυνσης μέχρι το τέλος του 2020, πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε τα αποτελέσματα μιας συνολικής ε, ανάλυσης έτσι ώστε ε, να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα κριτήρια και όλες οι μετρήσεις λαμβάνονται υπόψη. Ε, όσον αφορά τώρα τις, ε, τα επιτόκια χωρίς ε, κίνδυνο υπό το, την αφαιρεγγιότητα 2 λαμβάνονται υπόψη, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των επιτοκίων. Αυτές λαμβάνονται υπόψη, λέω, οι εκπτώσεις όσον αφορά τις ασφάλειες και τις επιβαρύνσεις τους η ΕΙΟΠΑ υπολογίζει στο, στα ε, επιτόκια και ε, έναν ε, διαφανή και προληπτικό τρόπο αντιμετώπισης που όμως θα βασίζεται οπωσδήποτε σε αντικειμενικά κριτήρια. Λαμβάνουμε υπόψη την ευρωπαϊκή αγορά κατανοούμε ότι οι προτινόμενες τροπολογίες στον κανονισμό έχουν ως στόχο ε, τη διασφάλιση συγκεκριμένων τροποποίησεων και αλλαγών όσον αφορά την μεθοδολογία υπολογισμού και ε, αυτό να γίνεται στο κατάλληλο επίπεδο. Ζητούμε να ληφθούν υπόψη και κάποια πρακτικά θέματα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν ε, ληφθεί υπόψη. Όσον αφορά τώρα ε, την προσαρμογή, ο υπολογισμός της προσαρμογής αυτής συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού ε, της αύξησης και των συγκεκριμένων προϋποθέσεων αναχώρα, των συγκεκριμένων προποθέσεων αναχώρα αναφέρονται λεπτομερώ στην οδηγία για την εφερεγγιότητα 2. Ε, η ΕΙΟΠΑ έχει άλλωστε σε ε, μηνιαία βάση ε, υπολογίσει και δημοσιοποιήσει ε, αυτούς τους υπολογισμούς με έναν τρόπο σόφρονα και διαφανή. Επίσης η ΕΟΠΑ έχει την δυνατότητα να υπολογίζει την συγκεκριμένη αύξηση αναχώρα καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τεχνικών λεπτομεριών όπως ας πούμε επιλογή των στοιχείων που θα οδηγήσουν στον ε, υπολογισμό. Να σας πω εν ε, συντομία και για να τελειώσω ότι η ΟΠΑ αυτή τη στιγμή αναλύει την εφαρμογή ε, της ε, προσαρμογής ως μέρος της αναδιάρθρωσης των μακροχρόνιων μέτρων διασφάλισης έτσι όπως απαιτεί ε, η οδηγία για την ε, αφαιρεγγιότητα 2 και θα δούμε πώς θα έχουν τα πράγματα τον Ιούνιο του 2020. Ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια μικρή αναθεώρηση προς το παρόν. Ναι. Θα δώσω το λόγο στους ομιλητές. Ο Μάρκος Φέμπερ από πλευράς του ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18 Σεπτεμβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου του 2018 ανέφερε ε, στην Επιτροπή τις ε, προτεραιότητες ε, που θεωρούμε πως ισχύουν σε ό,τι αφορά αυτή την επανεξέταση της οδηγίας. Καταρχήν, μείωση των κινδύνων, μετά προσαρμογή των, του υπολογισμού σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ε, ίδια κεφάλαια έτσι ώστε ακριβώς να υπάρξει καλύτερη συστοράκηση απέναντι σε κινδύνους και ε, τρίτον βέβαια η προσαρμογή της μεταβλητότητας. Ε, πέραν όμως μερικών μικροτροποποιήσεων σε ό,τι αφορά τα εργαλεία, σε ό,τι αφορά τα ίδια κεφάλαια, τίποτα δεν ελήφθη σε υπόψη στην στον του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα ήθελα να μου πείτε γιατί συνέβη αυτό αφού είχατε δεσμευθεί ότι θα λάβετε δεόντω υπόψει σα ε, τι ε, προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του review, στο πλαίσιο τη επαναξιολόγηση ε, και γνωρίζετε, συνειδητοποιείτε ότι έχει το δικαίωμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει ένα τέτοιο κατεξουσιοδότηση κανονισμό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχετικά εργαλεία για τα ίδια κεφάλαια, αποφασίσατε να μην ακολουθήσετε, όπω είπατε και στην παρουσίασή σα, μια προσέγγιση για το ring fencing, για την κλειστή διάρθρωση. Αλλά παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά αφορά το, τα, τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις υπάρχει ε, ε, συγκεκριμένη απέτηση σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ε, και ότι τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες επενδύσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Αυτή λοιπόν η ακαμψία αν θέλετε σε ό,τι αφορά το πλαίσιο ουσιαστικά οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα με εκείνο του ring fencing παρότι η ίδια, ο ίδιος ο όρος του ring fencing απουσιάζει πλέον από το ξεδόν του Άρα λοιπόν ε, η εφαρμογή αυτών των ε, διατάξεων ε, γίνεται δύσκολη και μη ελκυστική για τους επενδυτές και για, τους, για τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν αυτή η προσέγγιση που ακολουθείτε πράγματι θα, θα, διασφαλίσει την ελκυστικότητα αυτών των επενδύσεων σε, αυτές τις, σε αυτούς τους τομείς. από εκεί και μετά, τον Ιούνιο του 2017 ε, είχε ε, προβεί σε μια τροποποίηση του σχετικού του κανονισμού ε, στο ε, πλαίσιο της οδηγίας της Φερεγγιότητας 2 ε, ακριβώ επειδή ήθελε να καταστήσει τι επενδύσει σε υποδομέ σε πιο ελκυστικέ. Μπορείτε λοιπόν να μα πείτε ότι πράγματι στέφθηκε με επιτυχία αυτή η προσπάθεια που κάνατε. Δηλαδή υπήρξε αύξηση των επενδύσεων στι υποδομέ. Και μας είπατε τώρα πόσο σας ενδιαφέρει πάρα πολύ η αξιολόγηση του 2020. Θα ήθελα όμως να ακούσω από εσάς ποιες είναι οι προτεραιότητες τις οποίες έχετε θέσει σε το πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης. Εγώ να θέσω τρία σημεία εδώ. Περισσότερη αναλογικότητα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων και την ε, ε, ε δημοσίευση ιδιωτικών στοιχείων, δηλαδή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη περισσότερο η, ε, ε, αρχή της αναλογικότητας και για παράδειγμα λαμβάνοντας υπόψη και εκείνο που είχαμε προβλέψει σε ό,τι αφορά τις μικρότερες τράπεζες. Μετά, το δεύτερο στοιχείο ότι θα πρέπει η εποπτεία και η γενικότερη εξέταση των κινδύνων θα πρέπει να προσανατολίζεται εξατομικευμένα ακριβώς το προφίλ κινδύνου της, της κάθε τράπεζας, του κάθε επενδυτή και μετά θα πρέπει ε, ω τρίτο στοιχείο να ε, προβλέψουμε ε, ένα πλαίσιο σε ό,τι αφορά και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές και όχι μόνο βραχυπρόθεσμη λύση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ποιος θα απαντήσει και οι δυο σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ευχαριστώ. Όσον αφορά τις προτεραιότητές μας για την αναθεώρηση του 2020, είναι κάπως νωρίς να πούμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε πάντως είναι να έχουμε μια ευρή αναθεώρηση προκειμένου να μην αφήσουμε κανένα σημαντικό θέμα στην πάντα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε κάνει και μια ευρία έκκληση για βοήθεια από την ΕΙΟΠΑ, για συμβουλές από την ΕΙΟΠΑ. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και που είναι και στην καρδιά της αναθεώρησης είναι αναθεώρηση του πακέτου για τις μακροχρόνιες εγγύσεις. Γιατί όπως ξέρετε ήταν και το αντικείμενο περίπλοκων συζητήσεων εδώ. Οπότε αυτό σίγουρα είναι μια προτεραιότητα για μας. Κατά τα άλλα, θέλουμε να δούμε τι θα βγει από τις συμβουλές που θα μας στείλει η ΟΠΑ και τι θα βγει και από τις διαβουλεύσεις που θα κάνουμε και μετά θα αποφασίσουμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητές μας ε, αντλώντας μαθήματα από τη διαδικασία αυτή. Βέβαια σημείωσα τις προτεραιότητες που ανέφερε ο κύριος Φέρμπερ. Τώρα έρχομαι στα τρία στοιχεία κλειδί που ανέφερε ακριβώς ο κύριος Φέρμπερ. και τα οποία περιλαμβάνονται και στην επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σας τα πω με τη σειρά 1-1. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το περιθώριο κινδύνου. Εδώ επικεντρωνόμαστε κυρίως στο κόστος του κεφαλαίου, που έχει μεγάλη σημασία για τον υπολογισμό του περιθωρίου κινδύνου. Η ΕΟΠΑ έκανε μια ποσοτική ανάλυση σε βάθος, χωρίς προκαταλήψεις, όσον αφορά ε, το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η ΟΠΑ είναι ότι το κόστος του κεφαλαίου είναι στην πραγματικότητα υψηλότερο από το 6%. Και γι' αυτό η ΟΠΑ σύστησε να μείνουμε στο 6% που έχουμε τώρα και να μην αυξήσουμε το κόστος ε, κεφαλαίου και το περιθώριο κινδύνου κάποιοι θεωρούν ότι είναι καλό το ότι σταθεροποιείται το καθεστώς. Συμφωνούμε βέβαια ότι ο σχεδιασμός του περιθωρίου κινδύνου θα έπρεπε να αναθεωρηθεί εν ώψη του 2020 και γι' αυτό ζητήσαμε από τον ΙΟΠΑ να αναθεωρήσει σε αυτά τα πλαίσια, με τη Solvency 2 δηλαδή, το περιθώριο αυτό κινδύνου. για τις μακροχρόνιες μετοχικές επενδύσεις. Εδώ κάναμε πολλά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε διάφορες πλευρές προκειμένου να διευκολύνουμε ήδη από τώρα. Ε, αρχίσαμε με αναθεωρήσεις που κάνουμε όσον αφορά τις επενδύσεις σε μετοχές, περιμένοντας βέβαια την ευρύτερη αναθεώρηση του 2020. Δείξαμε επίσης ότι ακούσαμε και τους ε, ενδιαφερόμενους μετά την παρουσίαση του πρώτου σχεδίου μας και μειώσαμε την απέτηση από 12 σε 5 χρόνια για διακράτηση και έχουμε επίσης μειώσει και την αναφορά στο ring fencing την κλειστή διάρθρωση. Εδώ βέβαια θα έπρεπε να βρούμε μια καλή ισορροπία ανάμεσα στους στόχους EFSMU και την επιθυμία που έχουμε να προωθήσουμε τις μετοχικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία εκείνων που διακρατούν τέτοιες ε, επενδύσεις. Βέβαια, είναι θέμα συμβιβασμού στον οποίο θα καταλήξουμε. Με την περίοδο των πέντε ετών πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στο πιο χαμηλό επίπεδο αυτού που θεωρείται μακροχρόνιο. Και ήταν πολύ σημαντικό για μας οι ασφαλιστικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τις μεταχικές επενδύσεις για να καλύπτουν απώλειες που έχουν αλλού στον ισολογισμό τους. Αυτό για μας ήταν πολύ βασικό για την προστασία των ε, αποταμιευτών. Τώρα το θέμα της προσαρμογής της μεταβλητότητας. Εδώ η ανάλυση μας ήταν ότι οι αλλαγές στην συνιστόσα ε, χώρας πρέπει να γίνεται στο πρώτο επίπεδο από τον νομοθέτη. Και αυτό ακριβώς είναι που αποφάσισε να κάνει ο νομοθέτης. Βέβαια συμφωνήσαμε ότι πρέπει να δούμε ευρύτερα το θέμα της προσαρμογής μεταβλητότητας για να διασφαλίσουμε ότι στην πράξη λειτουργεί ικανοποιητικά και για όλες τις χώρες. Και σίγουρα αυτό σχεδιάζουμε να κάνουμε στα πλαίσια της αναθεώρησης του 2020. Αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εκ μέρους τη ΕΙΟΠΑ τώρα. Θέλετε κι εσείς να σχολιάσετε παρακαλώ. Επιτρέψτε μου κι εγώ να επανέλθω στο τελευταίο που ακούσαμε για την αναλογικότητα και τις προτεραιότητές μας που θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όντως θα συμπεριληφθούν στα θέματα που μας έδωσε για αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε για την αναλλαγικότητα σίγουρα είναι ένα συγκεκριμένο θέμα που εντοπίζεται στις αναφορές που γίνονται για την ενημέρωση. Υπάρχουν αυτά τα θέματα και στις απαιτήσει για, την ενημέρωση και θα παραμείνουν και στην αναθεώρηση του 2020. Τώρα, για την ε, προληπτική εποπτεία για την ελευθερία εγκατάσταση και ποια είναι η πιο σωστή θέση και αυτό περιλαμβάνεται στην αναθεώρηση του 2020 και οι μακροχρόνιες μετοχικές επενδύσεις βάσει των όσων είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα, εδώ ζητούμε μια πλήρη ανάλυση για τη μεταχείριση των μετοχικών επενδύσεων και είναι και αυτό κάτι το οποίο θα κάνουμε. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των σοσιαλιστών τώρα, θα ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι η ισορροπία της πρότασης τροποποίησης της τροποποιημένης πράξης δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό, ούτε και το θέμα της έγκαιρης ε, προειδοποίησης. Θα προχωρήσει σίγουρα αυτή η πράξη. Μια που πρόκειται για μια μικρή αναθεώρηση εν αναμονή της μεγάλης, έτσι. Πάντως πριν καταλαβαίνω ότι όπως συμβαίνει συχνά υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τον κλάδο για το πώς θα τεθούν σε εφαρμογή όλα αυτά από πλευράς ε, χρονοδιαγράμματος αυτή η αναθεώρηση κατά πόσο θα περιμένουμε το 2020, μήπως είναι καλύτερα να βάλουμε το 2021, έπειτα για τις ε, απαιτήσει αναφοράς, reporting και πόσο αυτό θα επηρεαστεί με τα όσα ήδη ισχύουν η κατεξουσδότηση πράξη σίγουρα θα επηρεάσει τις υποχρεώσεις reporting για το δεύτερο εξάμεινο. Δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να βοηθήσει όλους αυτούς ε, του κλάδου ή άλλους οι οποίοι μας ακούν και αναρωτιούνται. Ναι, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι περισσότερο ερώτηση, αλλά θέλω να πω και δύο λόγια για την μεγάλη αναθεώρηση. Υπάρχουν τρεις πτυχές που για μας είναι σημαντικό να λυθούν υπόψη. Και μια που εκφράζουμε ευχές για τους ανθρώπους που θα μας διαδεχτούν. το πρώτο θέμα είναι αυτό που είπατε κι εσείς, οι μακροχρόνιες ε, μετοχικές επενδύσεις. Πράγματι, ό,τι έχει γίνει με το hashtag και με τα κείμενα εφαρμογή. είτε πρόκειται για την ενημέρωση, είτε πρόκειται για το benchmark, είτε πρόκειται για ταξινόμηση, να συμπεριληφθούν στις μακροχρόνιες αυτές μετοχικές επενδύσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Φαντάζομαι ότι είναι ευαίσθητο θέμα. Το δεύτερο, επανέρχομαι στα εσωτερικά πρότυπα. Παρατηθήκαμε από αυτό το θέμα την τελευταία φορά και θέλω στις ρήτρες αναθεώρησης να συμπεριληφθούν και να γίνεται σαφώς ομνία το ότι θα πρέπει να καλύπτει η μεγάλη αναθεώρηση. Οπότε ρωτάω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα προετοιμάσει αυτή την πτυχή της μεγάλης αναθεώρησης. Γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται πιο ευάλωτη αν δεν προχωρήσει σε περισσότερη ολοκλήρωση όσον αφορά την εποπτεία των εσωτερικών μοντέλων στον κλάδο των ασφαλίσεων στην Ευρώπη. Μια που επιθέσεις ή τέλος πάντων έλλειψη επεξηγήσεων θα υπάρχει στη, είναι κάτι που θα υπάρχει στη διεθνή σκηνή και θα χρησιμοποιήσουν διάφορες εταιρείε που χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει πιο αποτελεσματικό έλεγχος των εσωτερικών ε, μοντέλων. Στην Ευρώπη πρέπει να ενισχύσουμε τη φωνή εκείνων που θέλουν να συνεχίσουν να μπορούν να υποφελούνται από τα εσωτερικά μοντέλα. Ναι, ξέρω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι περισσότερο ερωτήσει μου, αλλά και αν η ΟΠΑ θέλει να προσθέσει κάτι, ευχαρίστω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ για τα ενθαρρυντικά λόγια όσον αφορά ε, την ε, κατεξουσιοδότηση πράξη από το Κοινοβούλιο και την υποδοχή της δηλαδή από το Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε μια καλή ισορροπία στο κείμενο. Όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση του 2020. Οι εργασίες βεβαίως έχουν ήδη ξεκινήσει. Η ΕΙΟΠΑ επίσης και αυτή ε, προστρέχει. Το ε, θέμα βεβαίως θα ολοκληρωθεί το 19 και το 20. Ε, δεν πρέπει να ελπίζουμε νομοθετική πρόταση πριν από το τέλος 2020 γιατί η πρώτερη εργασία είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά την μελέτη αντικτύπου κυρίως που είναι περίπλοκη. Επομένως προς ώρας προβλέπουμε το νομοθετικό, την νομοθετική πρόταση στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 για να έχουμε αρκετό χρόνο έτσι ώστε να δουλέψουμε όλα τα περίπλοκα ζητήματα τα οποία προκύπτουν ε, όσον αφορά το reporting την υποβολή αναφορών εκθέσεων. Η ημερομηνία εφαρμογής θα εξαρτηθεί από την περίοδο ελέγχου και εξέταση από τον νομοθέτη. Εν τω μεταξύ το κείμενο έχει ήδη δημοσιευθεί, είναι ήδη ε, γνωστό, ε, το γνωρίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες μπορούν να προετοιμαστούν. Και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι στην ουσία τα reporting templates δεν αλλάζουν. Ε, αυτά θα τροποποιηθούν σε ένα τεχνικό πρότυπο εκτέλεσης αργότερα. Τέλος, όσον αφορά τα εσωτερικά ε, μοντέλα, όπως είπατε, ε, αυτό αυτό το σημείο αφορά την τελική αναθεώρηση του 2020. Οπωσδήποτε δεν το παραβλέπουμε το θέμα αυτό και συμφωνούμε με εσά ότι θα πρέπει σε διεθνές επίπεδο να είμαστε σε θέση να δείξουμε ότι έχουμε ισχυρά εσωτερικά μοντέλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θυμόμαστε και τα προβλήματα που είχαμε όσον αφορά αυτά τα μοντέλα στον τραπεζικό κλάδο και δεν θέλουμε να επαναληφθούν τα προβλήματα αυτά. Άρα μα απασχολούν στην Κομισιόν. Δεν θέλω να σας πω ακριβώς τι θα κάνουμε, γιατί πριν από μερικές μέρες ε, έγιναν δεκτά τα πρότυπα ΣΥΖΑ και επομένως οπωσδήποτε μπορώ να πω ότι μπορεί να βελτιωθεί ε, το κείμενο. Ε, πρόεδρος, τουλάχιστον κατανοείτε και εσείς ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά το πρασίνισμα, το greening ε, του τομέα των ασφαλιών. Έχετε να μας πείτε κάτι. Ναι, όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, η ΕΙΟΠΑ ήδη εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό και θα αποτελέσει οπωσδήποτε και ένα από τα στοιχεία αναθεώρησης του 2020. Ε, δεν ξέρω αν ο κύριος Φέρμπερ θέλει να πει κάτι. Όχι, δεν βλέπω άλλους συναδέλφους. Ε, εκπρόσωπος ΕΙΟΠΑ, ναι. Ναι. Όσον αφορά αυτό που εσείς ονομάζετε ε, μεγάλη αναθεώρηση και το χρονοδιάγραμμα η ΕΙΟΠΑ, ε, πρώτο θα έχει την ε, γνωμοδότηση του Ιουνίου 2020. Βεβαίως θα προχωρήσουμε μέσω διαβουλευτικής διαδικασίας ε, επί της γνωμοδοτήσεως και αυτό θα λάβει χώρα το τελευταίο τρίμηνο αυτού του έτους. Όσον αφορά ε, το reporting και την ε, ε, επιρροή επί του reporting της της πράξης θα προταθούν κάποιες τροπολογίες με την προϋπόθεση βεβαίως ε, και με την επιφύλαξη μάλλον ότι δεν, έχει ολοκληρωθεί, ε, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες ε, και που, με, το, με την προϋπόθεση ότι ενδεχομένως θα υπάρχει αρκετός χρόνος. Επίσης και η ταξινόμηση είναι σημαντική και θα ληφθεί η υπόψη και αυτή στις τροπολογίες και στην διαβούλευση της 1ης Ιουνίου που θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες προσχέδιο των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων ε, μέχρι τον Ιούλιο. Και βεβαίως θα ακολουθήσουμε ε, και την πορεία που είχαμε ακολουθήσει και με τις προηγούμενες ε, τροπολογίες για το reporting. Τέλος, όσον αφορά το πρασίνισμα των ασφαλείο, του ασφαλιστικού τομέα, μια πρώτη υπαρχή συμβουλών όσον αφορά τους κινδύνους ε, της βιωσιμότητας ε, μέχρι το καλοκαίρι και ε, συμπερίληψη στο Solvency 2, στη 2 των στοιχείων αυτών μέχρι το Σεπτέμβριο του 19. και τουλάχιστον ε, σας έχει δοθεί και πλήρης εντολή για τα θέματα αυτά. Πολύ ωραία. 25 ε, χρόνια έχω σε αυτό το σώμα και μάλιστα τότε η ΕΚΟΝ λεγόταν ΕΜΑΚ αλλά σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα στην ΕΚΟΝ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ολοκληρώνω λοιπόν αυτήν την δουλειά ε, με την συζήτηση της ε, κατεξουσιοδότηση πράξης ε, για τη Φερεγγιότητα 2. Είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να τελειώσουμε και να κλείσουμε την περίοδο με αυτόν τον τρόπο. Να σας πω ότι ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά ε, που συμμετείχα σε εργασίες αυτής της Επιτροπής και ελπίζω ότι οι συνεχιστές του έργου μας θα είναι εξίσου δεσμευμένοι και στρατευμένοι με εμάς. Ευχαριστώ πολύ.